Yeah. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Συνεχίζουμε με τις εργασίες Επιτροπής μας. Περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Ώρα των ερωτήσεων σχετικά με τον κανονισμό του ΡΙΤΣ. Το μεγάλο αυτό πακέτο της τελευταίας θητείας, το οποίο εντωμεταξύ βρίσκεται στη φάση της εφαρμογής. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα στο κοινό και οι συνάδελφοι εκμεταλλεύτηκαν την ε, ευκαιρία να θέσουν μια σειρά ερωτημάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζω τον κύριο Χάιντς Τσούρεκ, τον ε, Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς ήρθατε. Και δίπλα του είναι ο κύριος Γκους Μποσάρτ, διευθυντής ε, χημικών των υδάτων και της βιοτεχνολογίας. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Σκεφτήκαμε να χωρίσουμε τα πολλά ερωτήματα σε τρεις ομάδες εδώ πέρα. Το ένα αφορά την καταγραφή, την υπηρεσία καταγραφής και τα τέλη. Δεύτερον, λίστα υποψηφίων ουσιών παράρτημα 14 και 13. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε και πολλά πράγματα, ειδικά οι καινούργια, αλλά θα ακούσουμε οπωσδήποτε τι είναι. Και το μπλοκ 3 αφορά επίδοση ποινών, πειράματα σε ζώα, αντίκτυπος του ρίτς, σχέσεις ε, με την άλλη νομοθεσία, με λυπή νομοθεσία και νανοηλικά. Αυτές οι τρεις ομάδες προτείνω να ακούσουμε πρώτα τον ε, κύριο Γενικό Διευθυντή και μετά να περάσουμε στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για το που βρίσκεται η εφαρμογή του ΡΙΤΣ και θα ήθελα να πω αμέσως πως ε, κάποιες ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν μόνο από την Κομισιόν γιατί δεν είναι μόνο δική μας αρμοδιότητα γιατί το ΡΙΤΣ όπως ξέρετε είναι ένα μεγάλο δίκτυο και απαιτεί συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων και η Κομισιόν είναι ένας από αυτούς. Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του συναδέλφου του Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος γιατί βρίσκεται στο Μπανκόκ για να προετοιμάσει τη διάσκεψη της Κοπενχάγης. Και νομίζω ότι εκεί είναι πιο επίγουσα η παρουσία του και απαραίτητη από ότι εδώ και κατά τα λοιπά έχω να κάνω την εξής πρόταση κατά, τις, κατά τη διάρκεια των απαντήσεων των ερετήσεων που μας έχετε αποστείλει και γραπτός θα είμαι κάπως πιο αναλυτικός για να βοηθήσω και τους νέους βουλευτές που δεν ήταν εδώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης του ΡΙΤΣ για να τοποθετηθούμε σε κάποιους ε, ειδικούς τομείς του Ρίτσι. Αν ε, συμφωνείτε να περάσω σε μια σύντομη γενική παρουσίαση και μετά να περάσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα με τα μπλοκ όπως προτείνατε εσείς. Έχουμε μέχρι τις 11 η ώρα λέει ο κύριος Λάινεν οπότε μία ώρα και ένα τέταρτο, αλλά ας ε, ξεκινήσουμε. Πείτε μας πρώτα απ' όλα πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Θα το κάνω για να είμαστε τις πιο απλοί στην γνωστή γλώσσα της Κομισιόν, δηλαδή τα άσχημα αγγλικά. Uh, Χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να σας μιλήσω σε αυτή τη φάση εφαρμογής του <clears throat> προγράμματος. Rich είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα νομοθετήματα τα οποία έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ε, πρώτη θητεία του Πρόεδρου Μπαρόσο και του προηγούμενου Κοινοβουλίου και κάνει την Ευρώπη όλο αυτό να είναι μια ηγέτη στα θέματα κανονιστικού πλαισίου για, τα, για τις χημικές ουσίες. Επιδιώκει πολλά πράγματα συγχρόνως στο ΡΙΤΣ, προστασία της ανθρώπινης υγείας, προστασία του περιβάλλοντος, πρόθεση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμασίας, ελεύθερη κυκλοφορία χημικών ουσιών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας καθώς και της καινοτομίας στην χημική βιομηχανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει ένα κομβικό ρόλο στο να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει σωστή ισορροπία σε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο μεταξύ καταρχήν της προστασίας δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας και της πρόθεση της καινοτομίας από την άλλη πλευρά. Ο εισηγητής σας, ο κύριος Σακώνη, έγραψε ένα βιβλίο για την έγκριση του Ρίτς με δεύτερο τίτλο λέγοντας ότι ήταν πραγματικά ένα πολιτικό επίτευγμα η έγκριση του Ρίτς και συμφωνούμε με εμείς. Όλα αυτά ήταν μια ιστορική αναδρομή, αλλά αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει είναι τι γίνεται στην πράξη. Όπως είπα προηγουμένως, Είμαστε μόνο ένας από τους παίκτες μέσα σε εισαγωγικά που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του REACH. Η πιο σημαντική κινητήρια δύναμη πίσω από το REACH είναι ο φορέας για τις χημικές ουσίες που ήδη λειτουργεί, αλλά λειτουργεί κυρίως για την συγκεντρωτική διαδικασία έγκρισης. Τα κράτη-μέλη και οι αρχές τους όμως αντιμετωπίζουν δύο φορές το κάθε θέμα Αφενό με συνεργασία με τον κεντρικό αυτό φορέα και δεύτερον μέσω των διαδικασιών εφαρμογή στο εθνικό Έδαφο. Και έχουν και την ευθύνη για τις ουσίες του ΡΙΤΣ και για τους κινδύνους που επέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε και τη συνεργασία των βιομηχανικών κλάδων και των εμπλεκομένων που θέλουν να προωθήσουν την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών. Η πρώτη λοιπόν πρόκληση έχει αντιμετωπιστεί. Ήταν η δημιουργία του φορέα αυτού για τις χημικές ουσίες και ξέρετε ότι αυτό ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Γιατί χρειάστηκε να γίνει μέσα σε ένα πολύ στενό χρονικό πλαίσιο. Χρειάστηκε τεράστια αποφασιστικότητα από όλου αυτούς οι οποίοι πήγαν στο Ελσίνκι στα πλαίσια της δημιουργίας αυτού του φορέα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό το φορέα Ελπίζουμε ότι το... ο φορέας αυτός, ο οποίος δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2007, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή. Έχει 350 υπαλλήλου. Το 2010 όμως θα είναι το αποφασιστικό έτος, γιατί τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής με την πρώτη προθεσμία καταγραφής και θα έχουν τότε ένα τιτάνιο έργο να διεκπαιρεώσουν ως φορέας για τις χημικές ουσίες και επομένως θα χρειαστούν και περισσότερο προσωπικό φορέας αυτός μέχρι το 2010 θα παραμείνει εξαρτημένος από κοινοτικές επιδοτήσεις. Γιατί μόνο προς το τέλος του 2010 περιμένουμε από τα συλλεγόμενα τέλη να υπάρχει χρηματοδότηση αυτού του οργανισμού. Ξέρετε ότι η καταληκτική προθεσμία είναι το τέλος του Νοεμβρίου του 2010 και μόνο από τη στιγμή που καταγράφεται μια χημική ουσία τότε γίνεται και η τιμολόγηση και συλλέγονται τέλη. Επομένως μόνο προς το τέλος του 2010 θα αρχίσει ο οργανισμός αυτός να συλλέγει κονδύλια. Είναι επομένως απαραίτητο μέχρι τότε να υπάρχει μια επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν αρχικά. Και για μας ήταν το, η πρώτη σοβαρή δοκιμασία που χρειάστηκε να περάσει ο φορέας αυτός και ευτυχώς την πέρασε επιτυχώς γιατί υπήρξαν προκαταγραφές, προεγγραφές. που είχαμε εκτιμήσει σε κάποιο επίπεδο, αλλά το ο πραγματικός αριθμός ήταν 20 φορές μεγαλύτερος και μέχρι στιγμής έχουμε 2,7 εκατομμύρια εγγραφές, κάτι το οποίο μας ανάγκασε να αναβαθμίσουμε το μηχανογραφικό σύστημα του φορέα. Ακόμα και αυτό έγινε με επιτυχή τρόπο. Βλέπουμε τώρα ότι πέραν της πρώτης προθεσμίας καταληκτικής για την εγγραφή το Νοέμβριο του 2010. Υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική εφαρμογή νομοθετικής πράξης που είναι το νομοθέτημα για την ταξινόμηση συσκευασία και ετικετοθεσία των προϊόντων αυτών που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2011 και εκεί πάλι πάρα πολλέ εγγραφέ που έχουν αντιμετωπιστεί από το φορέα εμπλέκονται με, αυτή, με αυτό το νομοθέτημα. Το να δημιουργήσουμε λοιπόν και να συντηρήσουμε ένα μηχανογραφικό εργαλείο που θα κάνει όλα αυτά πραγματικότητα, το να δώσουμε κατευθυντήρε γραμμέ στη βιομηχανία, ιδίω στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά στον φορέα αυτό για τις χημικές ουσίες και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το φορέα αυτό. Λιγότερο από τρία χρόνια έχουν περάσει από την έγκριση της, του αρμόδιου κανονισμού, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στην πράξη έχουν επιτευχθεί οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Έχουμε λοιπόν το μηχανογραφικό σύστημα για το REACH, το οποίο παρέχει όλες τις υπηρεσίες που θέλαμε και από την αρχή του 2009 η βιομηχανία χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο για την ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εταιριών που παράγουν παρόμοιες ουσίες και επομένως για τον, ε, για τον υπάρχουν κοινά δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν ιστοσελίδα που περιέχει στοιχεία σε όλες τις κοινωτικές γλώσσες με απλό και ευσύνοπτο τρόπο. Υπάρχουν και ορισμένα παρατήματα του κανονισμού REACH τα οποία έχουν ε, αναθεωρηθεί και όπου διευκρινίζεται σαφώς ποιες είναι οι ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα παρατήματα 4 και 5, διευκρινίζοντας επίσης τις προϋποθέσεις για το, την εγγραφή στο παράτημα 11 και ανασκευάζοντας τα κριτήρια για την εγγραφή στο κεφάλαιο στο παράτημα 13. Και επίσης για τις δηλαδή ε, επίμονες βιοσορευτικές και τοξικές ουσίες. Τα πρώτα βήματα λοιπόν στην διαδικασία έγκρισης έχουν γίνει με την δημοσίευση του πρώτου υποψήφιου καταλόγου το 2008 και με τη συμπερίληψη ουσιών που θα πρέπει κατά προτεραιότητα να τύχουν εγγραφής. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε όμως ότι η μεγαλύτερη πρόκληση του ΡΙΣ δεν είναι για, την, ε, τον φορέα χημικών ουσιών ή για την Κομισιόν, αλλά για την βιομηχανία, η οποία θα πρέπει να διαμοιραστεί πληροφορίες για χιλιάδες ουσίες, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη πρόσθετων δοκιμασιών σε ζώα και να μην υπάρξει και πρόσθετο κόστος που θα επομισθούν. Θα πρέπει να γίνουν χιλιάδες αναλύσεις κινδύνου και να υποβληθούν αιτήσει εγγραφή και θα πρέπει να πληρωθούν τα αντίστοιχα τέλη από τη βιομηχανία. Πέραν λοιπόν του οικονομικού βάρους υπάρχει και τεράστια πρόκληση σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση και οι κύριοι φορείς της συνεργάζονται με την Υπηρεσία Χημικών Ουσιών και την Κομισιόν για να εξασφαλίσουν ότι καλύπτονται οι ανάγκες του βιομηχανικού αυτού κλάδου. Επίσης έχουμε εφαρμόσει ένα εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και την ετικετοθεσία για τις χημικές ουσίες. Με την ε, έγκριση και του ΡΙΤΣ και του νομοθετήματος για την ετικετοθεσία και την ταξινόμηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδειξε ότι μπορεί να είναι ηγέτη στην ασφαλή χρησιμοποίηση χημικών ουσιών. Κάποιοι ε, εταίροι μας έχουν διατυπώσει αμφιβολίες σε σχέση με το διεθνή αντίκτυπο του REACH, άλλοι βλέπουν πιο θετικά το θέμα αυτό και θεωρούν ότι υπάρχουν δυνατότητες να, να ευθυγραμμιστεί η δική τους νομοθεσία με το ΡΙΣ και να χρησιμοποιήσουν την νομοθεσία μας για την ταξινόμηση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών ως υπόδειγμα για να προχωρήσουμε σε ένα διεθνές σύστημα για τις χημικές ουσίες. Εμείς χαιρετίζουμε τα θετικά μηνύματα που έρχονται από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ όπου αναπτύσσουν αρχές για τη διαχείριση των χημικών ουσιών που είναι παρόμοιε με τις Ευρωπαϊκή Ένωση και σιγά σιγά συμμερίζονται την άποψη ότι μπορεί να θεωρηθεί ω υπόδειγμα η διαδικασία του ΡΙΤΣ και για αυτού. Επομένω, θέτουμε ένα παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα benchmark σε παγκόσμιο επίπεδο με το ΡΙΤΣ και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν την δραστηριότητα. Πολλά λοιπόν έχουν γίνει, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και είμαστε ε, σίγουροι ότι αν συνεργαστούμε όλοι θα μπορέσουμε να τι αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο να αναφερθώ στα θέματα αυτά και ο κύριος Μπόχομ είναι αυτός ο οποίος θα απαντήσει στα ερωτήματά σας όπως τις έχετε ομαδοποιήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για αυτούς οι οποίοι είναι καινούργοι στην Επιτροπή μας και δεν γνωρίζουν τα θέματα αυτά, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ χρήσιμα. Σας παρακαλώ έχετε το λόγο. Τώρα, όσον αφορά την απάντηση αυτών των πολλών και εξειδικευμένων ερωτήσεων, ε, θα ήθελα να απαντήσω. Έχουμε κάνει τη συνολική τώρα απάντηση. Πάμε αμέσω. Λίγη υπομονή δεν κάνει κακό. Ερχόμαστε στο πρώτο μπλοκ ερωτήσεων. Ξεκινάμε με τα ερωτήματα του κυρίου Ζέμπερ και Ρούλη και τα άλλα ερωτήματα για τα τέλη. Ίσως θα θέλατε να απαντήσετε. Νομίζω η διαδικασία είναι ότι ο ερωτών έχει το πρώτο δικαίωμα να θέσει ερώτημα και μετά μπορούν να επανέλθουν και άλλοι συνάδελφοι να συμπληρώσουν την προβληματική. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όσον αφορά την ε, εγγραφή, ήδη αναφέρατε τα μέλη του Κοινοβουλίου που έθεσαν τις ερωτήσεις αυτές. Να προσθέσω όμως και κάποιες ερωτήσεις για την προεγγραφή. Ε, ε, ερωτήματα τα οποία τέθησαν από τον κύριο Λάιεν, Λάινεν, τον αξιότιμο πρόεδρο της Επιτροπής. Ξεκινώ λοιπόν από τις ε, ερωτήσεις του πρόεδρου για το θέμα. για να μπορέσουν οι εταιρείε να ανταλλάσσουν στοιχεία, έτσι ώστε να αποφύγουμε μη αναγκαία πειράματα σε ζώα, το REACH ζητά από τις εταιρείε να προβούν ε, σε προεγραφή μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2008. Εν ώψη της σημασίας αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μαζί με ε, το ΕΚΑ, τα κράτη-μέλη και τις οργανώσεις ε, των κρατών μελών, της βιομηχανίας, ξεκίνησαν μια εκστρατεία για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση, η ενημέρωση και να ενθαρρυνθούν οι εταιρείε να προβούν στην προεγραφή. Μέχρι την προθεσμία αυτή, 2,75 εκατομμύρια προεγραφών αφορούσαν 143.000 ουσίες ε, και είχαν υποβληθεί από 65.000 εταιρείες. Ε, αυτό υπερεύει σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές, ε, ε, τους αρχικούς υπολογισμούς της Επιτροπής. Δημιουργήθηκαν ανησυχίες για τον αριθμό των εγγραφών που ε, θα μπορούσαμε να αναμένουμε μέχρι το τέλος της πρώτης προθεσμίας εγγραφής ε, ε, το 2010, την 31η Νοεμβρίου. Το ΕΚΑ, που είναι απευθεία υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της διαδικασίας εγγραφής, τώρα έχει αναλύσει τα στοιχεία της, που προκύπτουν από τα δεδομένα προεγγραφής και συνεργάστηκε με τη βιομηχανία για να αναπτύξει βελτιωμένους υπολογισμούς και εκτιμήσεις όσον αφορά τι εγγραφέ που θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2010. Ενώ να, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο βαθμό αβεβαιότητα, αυτέ οι βελτιωμένε εκτιμήσει δεν αποκλίνουν σημαντικά από τι αρχικέ εκτιμήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Το ΕΚΑ αναμένει ότι ο αριθμό των ουσιών θα ε, πλησιάζει τι αρχικέ εκτιμήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή γύρω σε 9.000. Επίσης, το ΕΚΑ θεωρεί ότι ε, οι εκτιμήσεις της Επιτροπής ως προς τον αριθμό των φακέλων εγγραφής, γύρω στις 25.000, εξακολουθεί να είναι κάτι το πιθανό. Αυτός ο αριθμός βεβαίως είναι περισσότερο αβέβαιος, παρόλο το ΕΚΑ πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε υπέρβαση ε, ε του αριθμού των 75.000 φακέλων. Τα αρχικά τέλη λοιπόν που θα μπορούσε να λάβει 2,7, ε, από 2,7 ε, εκατομμύρια εγγραφών δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντελώς αβάσιμο νούμερο. Βεβαίως βελτιώνουμε διαρκώς τις και Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τι εκτιμήσει αυτέ και τι εργασίε. Προ, προετοιμάζουμε επίση ε, προγραμματισμό επίγουσα ανάγκη για να αντιμετωπίσουμε πιθανή αιχμή στην εργασία. Ιδιαίτερα προβλέπεται 10.000 μεγαλύτερη ικανότητα για το σύστημα ταυτοποίηση του REACH από ό,τι περιμέναμε αρχικά. Επίση, προετοιμάζονται έκτακτα μέτρα τα οποία αφορούν του ανθρώπινου πόρου και ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού που συνήθω ασχολείται με άλλε ασχολίε, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να υποστηρίξουν την ομάδα εγγραφή κατά τι ε, περιόδου αιχμή, εάν βεβαίω προκύψει ανάγκη. Επιπροσθέτω, το ΕΚΑ ε, προβλέπει ε, και την πιθανότητα πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση. Αυτά όσον αφορά την προεγγραφή. Τώρα, ο κ. Ζήμπερ και Πρόντι έθεσαν ορισμένα ερωτήματα για την ίδια διαδικασία εγγραφής και θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω να απαντώ τα ερωτήματα αυτά. Η απάντηση είναι η εξή. Η διαδικασία εγγραφή, ε, όπω έχετε ε, ακούσει, έχει ξεκινήσει πλή, ε, πλήρω. Μέχρι στιγμή ε, έχουν υπάρξει μόνο ορισμένα προβλήματα και ο οργανισμό και η Επιτροπή παρακολουθούν την πρόοδο αυτή με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Με βάση τι πληροφορίε που παίρνουμε από τι οργανώσει του, κλάδου, είναι πιθανό οι εταιρείε να να, έχουν προλάβει και να γράψουν έγκαιρα τις ουσίες τους. Οι εγγραφές στα πλαίσια του ΡΙΤΣ ξεκίνησαν την 1η έκτου του 2008. Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί 120 εγγραφές περίπου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει δοθεί αριθμό εγγραφή και έχουν καταβληθεί ε, τα τιμολόγια. Γύρω, στα, γύρω στου 600 φακέλου εγγραφή ε, υποβλήθηκαν και η ποιότητα των ε, φακέλων βεβαίω θα πρέπει να βελτιωθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Οι ουσίε που, που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά εδώ και πολύ καιρό θα ενταχθούν στο σύστημα με τρία στάδια ανάλογα με το ποσό των χημικών ουσιών που παρασκευάζονται ή εισάγονται και με τις ιδιότητες των ουσιών αυτών. Η ε, βιομηχανία τώρα προετοιμάζει τους φακέλους εγγραφής για, την, το πρώτο στάδιο εγγραφής. Προθεσμία 30 Νοεμβρίου 2010. Ε, η ανταλλαγή δεδομένων για κάθε ε, για κάθε, περίπτωση γίνεται στα πλαίσια του SIFT, που είναι δηλαδή τα εσείς ε, τα φόρα ε, ανταλλαγής πληροφοριών. Ε, θα σας πω για άλλη μια φορά τι σημαίνει και μετά θα πω ΣΥΦ. φόρα ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες, ΣΥΦ όπου θα μπορούν να συμμετέχουν ε, όλοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και ο οργανισμό και οι οργανώσει ε, ε, του κλάδου και η Επιτροπή καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουν τι εταιρείε που αντιμετωπίζουν δυσκολίε ε, κατά την προετοιμασία των φακέλων εγγραφή. Ο οργανισμό και η Επιτροπή διοργάνωσαν και συμμετείχαν σε ένα αριθμό εργαστηρίων, συνδιασκέψεων και ε, άλλων φόρα για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα ΣΥΦ, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εμπλεκόμενοι να ε, ε, προβούν σε ανταλλαγή ερωτήσεων. Το θέμα ήταν πόσο χρόνο απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί ένα φάκελο. Ο μέσο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενό φακέλου είναι γύρω στον ένα χρόνο. Αλλά βεβαίως αυτό εξαρτάται από την ίδια την ουσία, ε, τους τόνους στους οποίους έχει κυκλοφορήσει και τη χρήση της. Σε ένα χρόνο ο ένα χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνει και τη συλλογή πληροφοριών και ε, πιθανά πειράματα, δοκιμέ και προετοιμασία του ίδιου του φακέλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ε, για τι ουσίε υψηλότερων όγκων μπορεί να απαιτηθούν δοκιμέ ε, που χρειάζονται και περισσότερο χρόνο. Δοκιμασίε που απαιτούν και περισσότερο χρόνο σύμφωνα με τα παρατήματα 9 και 10 του κανονισμού REACH. Αλλά τα, οι δοκιμασίε αυτέ δεν, δεν είναι απαραίτητο να διεξαχθούν πριν από την προθεσμία ε, εγγραφής. Γιατί στο, στον αρχικό φάκελο θα συμπεριλάβει προτάσεις για, τα, για τις δοκιμασίες. Τώρα, όταν δεν... Ε, η επεξεργασία των φακέλων ε, χρειάζεται ε, ένα μήνα περίπου, εάν δεν απαιτούνται δοκιμέ. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα, ο διοικητικό φόρτο θα αυξηθεί σημαντικά στην περίπτωση τη προετοιμασία μεγάλων κοινών υποβολών, όπου θα πρέπει να έχουμε το βασικό, εγγραφέ, το βασικό υπεύθυνο για την εγγραφή και ο οποίο θα αναφέρεται σε στοιχεία διαπραγματεύσει δεδομένων, ε, κατανομή του κόστου και τελικά συλλογή τη πληροφορία θα υποβληθεί κεντρικά. Αν επιτρέπετε τώρα, θα ασχοληθώ με το ζήτημα του κυρίου Πρόντι, με το ερώτημα του κυρίου Πρόντι, ο οποίο ε, αναφέρθηκε σε πιθανέ δυσκολίε ω προ την προθεσμία και στο κατά πόσο υπάρχουν απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει να συμμορφωθεί με το ΡΙΤΣ ή η χημική βιομηχανία. Η Επιτροπή δεν εξετάζει οποιαδήποτε αλλαγή στον κανονισμό όπως αναφέρεται, ο, γιατί ε, όσον αφορά τους βασικούς στόχους, καθώς επίσης ε, που παραμένουν αμετάβλητοι, καθώς επίσης και προσεκτικά εξεταζόμενος αντίκτυπος. Θα συνεχίσουν αυτές οι εταιρείε που θέλουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητε τους, πρέπει να συμμορφωθούν και να εγγραφούν έγκαιρα. Η Επιτροπή ε, όταν υπέβαλε την πρόταση αυτή εξέτασε εκτενώς τον αντίκτυπο του Ριτς και ιδιαίτερα ε, τον αντίκτυπο της εγγραφής στην διευρυμένη αξιολόγηση αντικτύπου. το, το συνεχιζόμενο κόστος και ο φόρτος εργασίας για την προετοιμασία των φακέλων, ε, οι εκτιμήσει αυτέ στηρίχθηκαν ε, σε ε, αυτά τα οποία υποστηρίζουν και οι ίδιοι οι επαγγελματίε. Η απέτηση για την εγγραφή νέων χημικών ουσιών ή οι λεγόμενε ουσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο phase-in, ξεκίνησε από την 1η Ιουνίου 2008 και εξή. Όσον αφορά τι ουσίε phase in, που ήδη υπήρχαν δηλαδή στην αγορά, ε, οι προθεσμίε εγγραφή εξαρτώνται από, την, ε, ε, ετήσια κυκλοφορία, από τον ετήσιο όγκο που παρασκευάζονται ή που εισάγονται και είναι 3,5 έω 11 χρόνια, ξεκινώντα από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού. Αυτό δίνει στη βιομηχανία τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμαστεί. Πρέπει επίση να μην ξεχνάμε ότι για του μεγάλου όγκου παραγωγή, οι χημικέ ουσίε που θα πρέπει να εγγραφούν μέχρι την 20 Νοεμβρίου 2010 για αυτέ τι ουσίε υπάρχουν ήδη πάρα πολλέ πληροφορίε. Όσον αφορά τώρα τον αριθμό των αναμενόμενων εγγραφών, δεν είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερο από τι εκτιμήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ε, διευρυμένη αξιολόγηση αντικτύπου από τα 2,75 εκατομμύρια προεγγραφών που, που έγιναν δεκτές, μόνο ένα σχετικά μικρός αριθμός θα καταλήξει σε πραγματική εγγραφή. Ο λόγος είναι ότι πολλές εταιρείες προέγραψαν σημαντικό αριθμό ε, χημικών, ουσίων, ε, χημικών ουσιών χωρίς να χρειάζεται αν θέλετε. Ε, προέρχονται από αυτές οι ουσίες, από γραφεία συμβούλων που αξιοποίησαν την ευκαιρία για να προσφέρουν τις υπηρεσίε τους στη χημική βιομηχανία. Οι εκπρόσωποι ε, ε, της βιομηχανίας που ήδη θεωρούν ότι είναι βασικοί υπεύθυνοι για την εγγραφή, δηλαδή προετοιμάζουν τις προεγγραφές εκπροσωπώντας εταιρείε που εμπορεύονται αυτές τις ουσίες επιβεβαιώνουν ότι μόλις 10% από τις εταιρείες που προέβησαν σε επαναγραφή έχουν την πρόθεση να εγγράψουν συνέχεια. Το οργανισμό, αλλά και η Επιτροπή όλοι κάνουμε κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουμε τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και όπως σας είπα, ο οργανισμό και η Επιτροπή συνδιοργάνωσαν διάφορες εκδηλώσεις για να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τα εργαλεία και την καθοδήγηση, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η Επιτροπή και ε, ο Οργανισμός προετοίμασαν και έδωσαν από τώρα ε, μεγάλο μέρος καθοδήγησης προς στη από τις πρώτες ημέρες του ΡΙΤΣ. Επίσης, οι οργανώσει του κλάδου βοήθησαν ιδιαίτερα και διευκόλυναν την εργασία των μελών του αναπτύσσοντας συγκεκριμένα ε, έντυπα και εργαλεία. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα εργαλεία, να σας πω ότι ο οργανισμός υποσχέθηκε να ε, δώσει το εργαλείο της ε, τεχνικής, ε, της τεχνικής ολοκλήρωσης, πληρότητας, μέχρι, έτσι ώστε, να το δώσει μέχρι τον Νοέμβριο, έτσι ώστε οι εταιρείε να μπορούν να, να είναι μέσα στην προθεσμία. Ε, επίσης, ε, για αρκετού μήνες υπάρχουν άλλα εργαλεία διαθέσιμα και των οποίων θα δοθεί η τελική έκδοση πολύ σύντομα. Να δώσω τώρα το, το λόγο στον συναδελφό μου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ να απαντήσω τα ερωτήματα τα δικά σας και του κυρίου Ζέμπερ για τη χρηματοδότηση των τελών ε, και την σύσταση της ε, υπηρεσίας του οργανισμού. Να το κάνω τώρα, αν και για την εμπειρία της σύσταση του οργανισμού θα πρότεινα να μιλήσετε και με τον κύριο Ντάντζιτς, τον διευθυντή του οργανισμού, ο οποίος οπωσδήποτε θα σας πει πολύ περισσότερα πράγματα για τις τρέχουσες δραστηριότητες. Ευχαριστώ όμως από την ε, εμπειρία μου ως ε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ε, εξ ονόματος να σας δώσω πληροφορίες οι οποίες θα είναι υπεύθυνε για τις τεχνικές ε, και οικονομικές πτυχές της κατάστασης του οργανισμού και για τη σύστασή του. Εάν ε, θέλετε και άλλες ε, πληροφορίες, να σας παραπέμψω στην έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού. Βλέπουμε πως ο οργανισμός συστάθηκε για να δώσει, να κάνει την καλύτερη δυνατή οικονομική και επιστημονική αξιολόγηση για τις χημικές ουσίες. Οπότε, ως εκ τούτου δεν πρόκειται μόνο για ένα μέσο που είναι κάπου συγκεντρωμένο, αλλά είναι και ένα δίκτυο διαφόρων επιτροπών σε όλα τα κράτη-μέλη και εμπειρογνωμών. Υπάρχουν διάφορε επιτροπές για τις οποίες μπορώ να πω ότι πρώτον έχουν συσταθεί και δεύτερον μπορώ να σα πω ότι έχουν επιτύχει μέχρι στιγμή. Υπάρχει η Επιτροπή για την Αξιολόγηση Κινδύνου και για τις ε, κοινωνικο-οικονομικές αναλύσεις που στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα στον οργανισμό να προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη στην Κομισιόν όταν μιλάμε για διαδικασίες αδειοδότησης και περιορισμού. Οι επιτροπές ε, των κρατών μελών που στόχο έχουν να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων αρχών στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή και το φόρουμ μετά που πρέ... θα είναι ένα δίκτυο στο οποίο οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα έρχονται σε επαφή με άλλους για την εφαρμογή του ΡΙΤΣ. Τα μέλη δε, της Επιτροπής ε, Αξιολόγησης Κινδύνου και Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης είναι εμπειρογνώμονες ε, που έχουν ε, πρόταθεί και οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και μάλιστα με βάση προτάσεις ε, ε, των κρατών μελών, οι οποίοι όμως είναι ανεξάρτητοι, δεν εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη, απλά ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την πρόταση των κρατών μελών. Επιλέγονται ή ορίζονται. η δεύτερη, πιο επιστημονική έτσι, κατεύθυνση της ε, Επιτροπής ή εκτός από αυτές τις επιστημονικές επιτροπές υπάρχει ένα φόρουμ που κατ' ουσίαν ε, συστάθηκε για να ανταλλάξουμε βέλτιστες διοικητικές πρακτικές ε, και εμπειρίες για τις στρατηγικές εφαρμογής. Και οι τρεις αυτές επιτροπές του οργανισμού στο φόρουμ ήδη από την αρχή του 2008 έχουν προχωρήσει στην σύστασή τους σε σώμα και εντωμεταξύ η Επιτροπή Ιράκ ε, Αξιολόγηση Κινδύνου έχει συνεδριάσει 7 φορές, η Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης 4 φορές, η Επιτροπή των Κρατών Μελών 8 φορές και το Φόρουμ 5 φορές. Επιπλέον ε, εντωμεταξύ υπάρχει μια πρώτη συνεργασία μεταξύ των Επιτροπών και του Φόρουμ έτσι ώστε κλείνει, να κλείνει αυτός ο κύκλος επικοινωνίας. Προσπαθήσαμε λοιπόν ε, μαζί με τον οργανισμό να διασφαλίσουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνία και διαφάνεια. Γι' αυτό αποφασίσαμε ότι όλα τα έγγραφα αυτών των ε, επιτροπών θα δημοσιεύονται κιόλας. στην ιστοσελίδα του οργανισμού για να τα βλέπει το κοινό. Και επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για διάφορες ομάδες συμφερόντων να λάβουν μέρο στην διαδικασία για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά τους και να μας πούν την άποψή τους. Και το φόρουμ αποφάσισε επίσης μία φορά το χρόνο τουλάχιστον να συμβουλεύετε τους ενδιαφερομένους με τον Πασκαλ. Μπορούμε λίγο να επιταχύνουμε, λέει ο κύριος Πρόεδρος. Αυτά ήταν υπό τον τίτλο «Σύσταση του οργανισμού». Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Κατά βάση υπάρχουν ε, τρεις ε, μέθοδοι, τρεις πηγές χρηματοδότησης του οργανισμού. Έχουμε μια κοινοτική επιδότηση. Δεύτερον, έχουμε τα τέλη από τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν ε, ουσίες. Και τρίτον, εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή κατ' ουσίαν εξαρτάται ο οργανισμός από την κοινοτική επιδότηση για το τέλος του έτους 2010, όταν θα αρχίσουν να εισραίουν τα έσοδα των τελών, υπολογίζουμε πως ε, θα κορυφωθεί αυτή η ροή το 2011 και μετά θα υπάρξει κάποιος χρόνος ε, μέχρι να μπορέσει να φτάσει ο οργανισμός να λειτουργεί χωρίς κοινοτική επιδότηση, αλλά νομίζω θα είναι εντός της θητείας αυτού του κοινοβουλίου. Θα μπορέσουμε μία μέρα να έρθουμε εδώ πέρα να ξαναζητήσουμε όμως κάποια κοινοτική επιδότηση γιατί μακροπρόθεσμα τα τέλη θα αρχίσουν να μειώνονται διαρκώς και θα χρειάζεται μια κοινοτική στήριξη, μια κοινοτική χρηματοδότηση και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι έχουμε την υποστήριξη της ε, Επιτροπής σας για την διάθεση μιας επιδότησης μέχρι το τέλος του 2010. Τώρα για το ερώτημά σας για το αν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα αυτό το μοντέλο. Όχι, αλλά δεν ήταν ποτέ αυτή η σύλληψη δηλαδή τα τέλη να χρηματοδοτούν όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σύντομοι, αλλιώς δεν θα προλάβουμε καθόλου. Έχουμε στον Ρίχα Τζέμπερ, αν θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για την ιδιαίτερα εκτενή παρουσίασή του. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα. Καταρχήν, από την έκθεση για το 2006 αναφέρθηκε ότι ο στόχος ήταν μια εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και υπήρχε τότε το γλωσσικό πρόβλημα. Από ό,τι ήξερα, οι πληροφορίε αρχικά ήταν μονάχα στα αγγλικά. Έχει καταφέρει πραγματικό Κομισιόν να παρουσιάσει τι πληροφορίε, ή μάλλον ο φορέα για τι χημικέ ουσίε, η ΕΚΑ, να παρουσιάσει την πληροφορία σε όλε τι κοινωτικέ γλώσσε. Καταλαβαίνω ότι αυτό σημαίνει και πρόσθετο κόστο μετάφραση, αλλά δεν είμαστε όλοι αγγλόφωνοι. <clears throat> και το δεύτερο ερώτημα. Αποφασίσαμε να προχωρήσει το πρόγραμμα REACH γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση για όλου και θα βοηθήσει και την ανθρώπινη υγεία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά και για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αλλά η Κομισιόν εξακολουθεί να παρακολουθεί ποιες είναι οι πρακτικές επιπτώσεις του REACH, τι εξοικονομήσεις προέρχονται από αυτό. Γνωρίζουμε κάτι καινούριο από όλα αυτά. Πώ προχωρούν τα πράγματα με τις αξιολογήσει αντικτύπου και τα λοιπά. Τι νέα στοιχεία έχει να μα δώσει για όλα αυτά η Κομισιόν δηλαδή. Παρακαλώ, σας παρακαλώ να είστε σύντομο, λέει ο πρόεδρο. <clears throat> Πρώτο ερώτημα, το γλωσσικό θέμα. Η πληροφορία είναι ε, διαθέσιμη με κάποια καθυστέρηση. Δηλαδή έχει επέλθει μια καθυστέρηση μέχρι τη στιγμή που μπορούν να δοθούν οι πληροφορίες σε περισσότερες γλώσσες από μονάχα από τα αγγλικά. Καταρχήν δινόντουσαν οι πληροφορίες μονάχα στα αγγλικά, αλλά σίγουρα αυτό προχωρεί και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε, αλλά φυσικά εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία, με την οποία οι πληροφορίες μας έρχονται και έχουν ελεγχθεί για να μπορέσουν να μεταφραστούν. Πρέπει να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και τότε μπορούν να τεθούν στη διάθεση όλων των επιχειρήσεων. Γιατί η βασική αρχή που διέπει την λειτουργία μας είναι να μην υπάρχουν σφάλματα, μετάφρασης ή οτιδήποτε άλλο μπορούσε να δώσει λαβή σε λαθασμένες πληροφορίες προς τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό έχουμε ένα σχετικά αυστηρό έλεγχο, ο οποίος βέβαια οδηγεί και σε κάποιες καθυστερήσεις. Πρέπει να εξασφαλίσουμε, πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι και ο φορέας για τις χημικές ε, ουσίες λόγω του υπερβολικού ίσως βάρους προεγγραφών είχε πράγματι πρόβλημα με το προσωπικό της, δεν είχε αρκετό προσωπικό για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα και επομένως θα ήταν απαραίτητο να έχει ο φορέας, μας, ο φορέας αυτός τις ικανότητες να μπορέσει να καλύψει την ε, απόσταση που έχει από την κατάσταση πλήρους ε, λειτουργίας. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Ήρθα κάπως καθυστερημένα γιατί ήμουν στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Έχω ένα ερώτημα τώρα προς την Κομισιόν. Είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλές προεγγραφές, 20 φορές περισσότερο από ό,τι περιμένατε. Είπατε ότι αυτό έχει και επιπτώσεις στο προσωπικό και την ανάγκη να υπάρξει στελέχωση με πρόσθετο προσωπικό στον φορέα αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και επίσης μήπως θα μπορούσε να γίνει κάτι με τις προθεσμίες, να ευκαμπτοποιηθούν κάπως οι προθεσμίες όταν έχετε τόσες πολλές προεγγραφές καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε, να σε όλες αυτές. Μήπως λοιπόν θα μπορούσε λόγω αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού εγγραφών μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλες αυτές τις ε, προεγγραφές και τις εγγραφές που θα έρθουν ή ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάποια αλλαγή ε, για να προσαρμοστείτε στις αιτήσει των επιχειρήσεων. Σύντομη απάντηση. Για τις ε, προθεσμίες δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, γιατί έχουν καθοριστεί και είναι απαράγραπτες. Αλλά αυτό το οποίο δεν θεωρούμε ιδιαίτερα πιθανό είναι ότι αυτός ο τεράστιος αριθμός των προεγγραφών θα επαναληφθεί και στο μέλλον. Δηλαδή δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει ένας τόσο μεγάλος αριθμός πραγματικών εγγραφών. Αλλά νομίζω ότι ήδη ο συνάδελφός μου απήντησε σε αυτό το ερώτημα. Για τις προθεσμίες πάντως νομικά δεν είναι δυνατό να τις αλλάξουμε. Ερχόμαστε ε, στα PPT, PPT τις ε, επίμονες, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες. Βέσλου, Λεπάζ, Ρόδο και Σλούτερ. Σας παρακαλώ να είστε και εκεί σύντομοι, γιατί έχουμε κάπως καθυστερήσει. Ευχαριστώ, θα κάνω ό,τι μπορώ. Μία ερώτηση που έκανε ο κύριος Σέμπερ για τις ε, πτυχές υγείας. Έχουμε κάνει μια βασική μελέτη, ξέρουμε ποιες είναι οι βάσεις ε, για την υγεία. Θα γίνει μια δεύτερη μελέτη, θα γίνει μετά η σύγκριση, οπότε η απάντηση είναι ναι πως συνεχίζουμε την έρευνα για τα ζητήματα υγείας και είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, για τις ανθεκτικές, βιοσυσορυφτικές και τοξικές ουσίες, Μιλάμε για επίμονες βιοσυσορευτικές και τοξικές ουσίες ή και άκρος ε, βιοσυσορευτικές και τοξικές. Ως, ε, μέλο, ως μέρος λοιπόν ε, της κοινή Αγγιστουρίτης αποφασίστηκε πώς θα πρέπει αυτά τα κριτήρια να επανεξεταστούν πριν από την 1η Δεκεμβρίου του 2008 για να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η διεθνή εμπειρία στην αναγνώριση τέτοιων ουσιών η Κομισιόν πράγματι οριστικοποίησε αυτή την εξέταση πριν τον Δεκέμβριο του 2008 και κατέληξε πως τα κριτήρια πρέπει να τροποποιηθούν. Η Κομισιόν θα οριστικοποιήσει την πρότασή της για την αλλαγή αυτών των κριτηρίων με βάση τα συμπεράσματα αυτής της αναθεώρησης. Στην πρόταση αυτή βεβαίως λαμβάνουμε πλήρως υπόψη τη συνεισφορά της δικής σας Επιτροπής αλλά και άλλων ενδιαφερομένων όσον αφορά την χρήση όλων των υπαρξών πληροφοριών για το πώς θα βρούμε αυτές τις ε, ανθεκτικές ισορρευτικές και τοξικές ουσίες και θεωρούμε πως το νομικό κείμενο του παρατήματος 13 θα πρέπει να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ουσίες χρησιμοποιώντας ε, μια στάθμιση ε, για να εφαρμόσουμε αυτά τα κριτήρια. Αναθεωρούμε αυτή τη στιγμή το σχέδιο κειμένου για να μπορέσει να υποβληθεί στην διαδικασία της επιτροπολογίας και να εκπληρώνει τον στόχο, δηλαδή να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η αποκτήσει εμπειρία. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον συνάδελφό μου, αν μου επιτρέπετε. Μετά από πέντε λεπτά θα τελειώσουμε, οπότε δυόμιση λεπτά έχετε. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για την συμπερίληψη ουσιών ε, υψηλής ανησυχίας στον ε, κατάλογο υποψηφίων. Να σας δώσω τις εξής πληροφορίες. Γνωρίζουμε τις ε, προσδοκίες διαφόρων για το ότι ο κατάλογος υποψηφίων θα πρέπει να αντανακλά την ανησυχία διαφόρων ενδιαφερομένων, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης τη λειτουργία του συστήματος. Οπότε προς στιγμήν συμφωνήσαμε να προτείνει μια πρώτη λίστα η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και ο οργανισμός και θα περάσουμε και σε μια δεύτερη λίστα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πως δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη με διαδικασίες που οι σε διαφορετικό πλαίσιο, σε νομοθεσία που προϋπήρχε του ΡΙΤΣ και πρέπει να έχουμε και έναν επαρκώς τεκμηριωμένο φάκελο. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές αρχές που θέλουμε να τηρήσουμε κατά την αξιολόγηση, γιατί το έργο αυτό για τη σύνταξη αυτού του καταλόγου είναι που πρέπει, είναι κάτι που θα πρέπει να μοιραστούμε με από όλους τους πιθανούς ενδιαφερομένους στον οργανισμό. Υπάρχει λοιπόν συνεχής διάλογος με όλους αυτούς του ενδιαφερομένους και το εξετάζουμε. Έχουμε λάβει και κάποιες πληροφορίες από κάποια κράτη-μέλη που έχουν κάνει κάποιες μελέτες και μας κοινοποιούν τα αποτελέσματα. Θέλουμε να μάθουμε ποια είναι αυτά. Θα σας κρατάσουμε λοιπόν ενήμερους για τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης και για τις προτάσεις που θα τεθούν μετά προς έγκριση από τον οργανισμό. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, ερωτήσεις για αυτά που ακούστηκαν. Σλούτερ. Ευχαριστώ. Είπατε ότι όσον αφορά τα κριτήρια για τα PBT αυτά θα λαμβάνετε υπόψη ε, τις απόψεις ε, των εμπλεκομένων στα κράτη-μέλη και των ενδιαφερμένων στα κράτη-μέλη. Και είναι σαφές ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη που εξέφρασαν άποψη ε, ακολούθησαν αυτή τη λύση που σημαίνει ότι θα συμπεριληφθούν και άλλε πληροφορίε όσον αφορά την ταυτοποίηση ε, σύμφωνα με τη Σύμβαση τη Στοκόλμη. Και δεν ξέρω, όταν λέτε τώρα. Γιατί κοιτάξτε, θα έπρεπε να έχετε κάνει αυτή την πρόταση από το Φεβρουάριο. Αυτό, ε, σε αυτό είχατε δεσμευτεί. Ε, δεν την είχαμε το Φεβρουάριο, τώρα είπατε ότι θα έρθει. Ε, αναρωτιέμαι πριν από το τέλο του χρόνου. Και μετά, το εξή όταν λέτε ότι ελήφθησαν υπόψη οι απόψει που, εκφρα... που εκφράστηκαν. Θα ακολουθήσετε δηλαδή τη λύση 3 που συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικές για τον εντοπισμό πέραν των βασικών κριτηρίων. Και συγγνώμη που θα είμαι κάπως περισσότερο επιστημονικός και ε, τεχνικός. Όσον αφορά τον ορισμό μιας βιοσορευτικής ουσίας, είναι ε, τα κριτήρια διαχωρισμού ε, οκτανόλης και ύδατος και ε, τα γενικά ε, κριτήρια είναι 100.000 ε, περισσότερα από τα γεγονότα. Τώρα είδαμε ότι αν η αναλογία είναι κάτω από τα 100.000 αλλά πάνω από 100 μπορεί να να, έχουμε γενικά ε, σωρευτικότητα, αλλά όχι στο νερό. Άρα λοιπόν πρέπει να διαβριθούν τα κριτήρια έτσι ώστε να δούμε και τη βιοσόρευση ε, στα, στους ανθρώπους ή στις ε, πολικές άρκτους που δεν ζουν στο νερό, αλλά παρόλα αυτά είναι βιοσορευτικές αυτές οι ουσίες. Τα νέα κριτήρια λοιπόν που προτείνεται θα λάβουν υπόψη αυτό το στοιχείο. Θα είναι σύμφωνα με την επιλογή 3, με τη λύση 3 και θα έχουμε τέλος πάντων την πρόταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχετε το λόγο σημαντικές και δύσκολες ερωτήσεις, Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Ναι, το καταλαβαίνουμε Δεν έχουμε κάπως καθυστερήσει. Σε ευχαριστώ που μας το επιθυμήσατε. Το ξέρουμε όμως και μας ανησυχεί, αλλά αυτό μας αποτελεί κίνητρο για να προχωρήσουμε και να σημειώσουμε πρόοδο. Είναι σημαντικό το θέμα. Κοιτάξτε, αυτό που θέλουμε είναι να λάβουμε υπόψη όλες τις πληροφορίες. Και αυτό καλύπτει και την δική σας την ερώτηση. Ναι, ξέρετε ότι είναι ευρύτερο ορισμός και γίνονται συζητήσεις. Αλλά πρέπει να δώσουμε και βεβαιότητα στι εταιρείε. Καταρχήν όμως θέλουμε να λάβουμε υπόψη, να είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνονται υπόψη όλες τις πληροφορίες. Θα θέλαμε να επανέλθουμε σύντομα με την πρότασή μας και να τα πούμε τότε, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε το γιατί μιλάμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάση, δεύτερη συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την απάντηση, αλλά δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε από τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί από τα μέλη της Επιτροπής μας σε σχέση με τον κατάλογο των υποψηφίων ε, ουσιών που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ότι έχει τύχει κάποια ερώτηση απαντήσεως πλήρους από την Κομισιόν. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε ότι έχετε το διάλογο αυτό με τους εμπλεκόμενους, αλλά πολλά κρατημέλη, τουλάχιστον ε, το γνωρίζει και η κυρία Βέστον και εγώ, έχουν ζητήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υπάρχουν πολλές ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες κτλ. Επίσης βιοσορευτικές κτλ. Όπου ισχύει μονάχα το 15 συν 15 που είναι αυτές οι ουσίες λοιπόν στον επίσημο κατάλογο. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για ένα από τους κύριους στόχους του ΡΙΤΣ, που θα μπορούσαμε να τον εξηγήσουμε καλύτερα στους απλούς καταναλωτές και που έχουν το δικαίωμα το ξέρουν. Λέει η νομοθεσία ότι ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να έχει μία απάντηση στο μαγαζί που αγοράζει παραγωγός χάρη οποιαδήποτε ουσία η οποία έχει εγγραφεί στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του ΡΙΤΣ για αυτό το προϊόν. Όταν όμως ο κατάλογος αυτός αποτελεί μονάχα ένα πολύ μικρό κλάσμα των ουσιών που επέχουν ειδική ανησυχία, τότε δεν πραγματοποιείται αυτή η αίτηση του καταναλωτή να ξέρει περί τίνος πρόκειται και έχουμε θέσει αυτό το ερώτημα στην Κομισιόν μέχρι ποια καταληκτική ημερομηνία πόσες ουσίες θα έχουν περιληφθεί στον κατάλογο αυτό και πώς θα γίνει η κατανομή καθηκόντων μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών για να επεκταθεί αυτός ο κατάλογος και εκεί πέρα δεν απαντήσετε. Φοβάμαι ότι μπορώ να απαντήσω. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να σας πω είναι... Μπορώ να σας πω ότι θα κάνει η Κομισιόν. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι μονάχα διαδικασία της Επιτρόπης, είναι μια κοινή διαδικασία και με τα κράτη-μέλη που βασίζεται και στην συμμετοχή των κρατών μελών. Εμείς ήδη ε, τον Ιανουάριο του 2009 κάναμε ένα κοινό εργαστήριο με τα κράτη-μέλη για να έχουμε μια κοινή βάση για αυτό το εγχείρημα και θέλουμε να συνενώσουμε τις προσπάθειές μας. Βάσει των συμπερασμάτων αυτού του εργαστηρίου, μια ομάδα από κράτη-μέλη ανέπτυξε μια προσέγγιση η οποία έχει σαν στόχο πρώτο να ταυτοποιηθούν οι ουσίες υψηλής ανησυχίας, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητος και επίσης να δημιουργηθεί εν καιρό ένας κατάλογος υποψηφίων ουσιών στα επόμενα χρόνια. Δεν θα είναι η μεγάλη έκρηξη λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε βάσει των προτεραιοτήτων να καταρτήσουμε αυτό τον κατάλογο. Το αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματο έχει παρουσιαστεί στα κράτη-μέλη, την ε, Κομισιόν και τον Φορέα Χημικών Ουσιών τον Ιούλιο και έχει συζητηθεί και στο Ελσίνκι τον προηγούμενο μήνα. Επομένως τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσουν ποια είναι η συνέχεια πρέπει να δοθεί σε αυτή τη δράση και μετά η επόμενη συνάντηση των αρμοδίων αρχών και για το ΡΙΤΣ και για τις μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες και τα λοιπά ουσίες θα πρέπει να επιληφθεί. Έχουμε αφήσει στα κράτη-μέλη που είναι οι κάτω χώρες, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία κτλ. να μας ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των δοκιμών τους και εμείς θα επιληφθούμε το θέμα του αυτού όταν γνωρίσουμε τι έχει επιτύχει η πρωτοβουλία αυτών των χωρών. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω δυστυχώς <clears throat> κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με τον αριθμό των ουσιών που εγγράφονται στον κατάλογο ουσιών υψηλής ανησυχίας. Μονάχα μπορώ να σας πω είναι ότι προσπαθούμε να λειτουργήσουμε όσο μπορούμε με πιο μεγάλη ταχύτητα για να έχουμε αυτόν τον κατάλογο το ταχύτερο δυνατό και να είναι όσο πλήρης μπορεί να είναι αυτός ο κατάλογος ανθρωπίνος βέβαια πάντα λέω. Παρακαλώ, κύριο Σλίτερ. Ευχαριστώ. Ε, είχε την καλοσύνη ο πρόεδρο να μου δώσει πέντε δευτερόλεπτα για follow-up στην ερώτησή μου. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο. Αλλά η, ε, η πολιτική είναι ιδιαίτερα απλή. Έχουμε 11 κράτη-μέλη, συν την Ορβηγία, συν τον Οργανισμό για τι χημικέ Ουσίε, που όλοι προτιμούν μια συγκεκριμένη επιλογή, όπω είπα πριν από λίγο. Συμπεριλαμβάνουν δηλαδή και άλλε πληροφορίε. Και μόνο δύο κατά. Το Ηνωμένο Βασίλειο και τη χημική βιομηχανία έχουμε τη Γενική ε, Διεύθυνση Περιβάλλοντος που θέλει την αλλαγή και την ε, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων που δεν τη θέλει. Ε, μήπως πρέπει να πάμε το θέμα στον Παρόζο και να πούμε ότι τώρα πρέπει να, να, παρα, παρακούσουμε την ε, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και να δούμε τι θέλουν τα κράτη-μέλη, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και να πούμε Ε, στον Εμένο Βασίλειο, συγγνώμη, χάσατε αυτή τη μάχη. Δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα και σας παρακαλώ να, να τελειώσετε πριν από το τέλος του χρόνου για να απλοποιήσετε αυτό το πολιτικό αγώνα. Έχουμε τόσα πράγματα να ασχοληθούμε αυτό το φθινόπωρο. Ε, μην ε, ε, κάνουμε λοιπόν και ανώφελες μάχες όταν η πλειοψηφία των κρατών και οι επιστήμονες είναι εξαιρετικά σαφείς. Ναι, πέντε δευτερόλεπτα, τα χρησιμοποίησατε σωστά, πολύ ωραία. Ε, αναγνωρίζετε το το ερώτημα και εν ευθέτω χρόνο θα το δείτε. Ε, δεν ήταν ερώτημα, ήταν μια έκκληση, τη σημείωσα. Θα το θέσετε στον Παρόσο λοιπόν. Ε, αν με ακούσει εμένα βεβαίως. Ωραία. Λέει ο πρόεδρος, στο δεύτερο μπλοκ είχαμε και το σημείο 6 μετά, ουσίες ε, προτεραιότητας και το παράρτημα 14, το ερώτημα των Ρόντε και Χάση. Θα τα απαντήσετε και αυτά. Ναι. Και εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση όπου σκοπεύουμε να δώσουμε μια σαφή και βέβαιη απάντηση σε όλους όσοι επηρεάζονται από αυτό και θέλουμε να υπάρξει μια καθοδήγηση. Ελπίζουμε να γίνει αυτό τις ερχόμενες εβδομάδες. Πριν το τέλος της εβδομάδας να υπάρχει πρώτα απ' όλα μια νομική βεβαιότητα και μετά να συντάξουμε αναλόγως και τις κατευθυντήριες γραμμές για να είναι διαθέσιμο το συντομότερο δυνατόν. Gibt's nachfragen? Να επανέλθετε στο ίδιο ερώτημα. Όχι. Περνάμε λοιπόν στο τρίτο μπλοκ. Ειδοποίηση, κοινοποίηση και ποινές. Ερώτημα Φερνάντες. Η απάντησή σας ποια είναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απάντηση είναι η εξής. Η εφαρμογή του ΡΙΤΣ είναι ευθύνη των κρατών μελών το άρθρο 125 υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να διατηρούν ένα σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων που θα ανταποκρίνει τις συνθήκες. Το άρθρο 126 προβλέπει πως τα κράτη-μέλη θα προβλέψουν ποινές απαραίτητες για παραβίαση του κανονισμού και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν τις θέσεις αυτές στην Κομισιόν πριν από το Δεκέμβριο του 2008 και κάποια, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή αμελητή. Κάποια κρατημέλη δεν έχουν ακόμα ειδοποιήσει την Κομισιόν όσον αφορά τις ποινές και το Δεκέμβριο του 2008 η Κομισιόν ξεκίνησε μία μελέτη για τα για τις ποινές ε, των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσει του ΡΙΤΣ. Θα σας δώσουμε λοιπόν μια γενική εικόνα και μια σύγκριση των διατάξεων ε, για την παραβίαση του κανονισμού. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα μετά κύριε Πρόεδρε. σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση της κινητοποίησης, τι έχει κάνει η Κομισιόν η Κομισιόν έχει ενημερώσει τα κράτη-μέλη για τις κοινοποιήσεις που λάβαμε το Δεκέμβριο του 2008 και τον Μάρτιο του 2009. Τον Ιανουάριο του 2009 η Κομισιόν απέστειλε μια επιστολή για να υπενθυμίσει τα κράτη-μέλη που δεν μας είχαν κοινοποίησει και, μας είπαν, και τους είπαμε πως ε, το να μας έχουν ε, κοινοποιήσει σημαίνει παραβίαση του ΡΙΤΣ και μπορεί να ξεκινήσουμε διαδικασία παραβάση και μάλιστα κινήσαμε διαδικασία παραβάση κατά των κρατών μελών αυτών. Οι επίσημες επιστολές ε, στάλησαν τον Μάιο του 2009. Τρίτο ερώτημα ήταν εάν η Κομισιόν έχει ήδη ειδοποιήσει κάποια κράτη-μέλη ε, ποιες ήταν οι δικαιολογίες ε, που ακούστηκαν. Δεν ακούστηκαν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι. Τα περισσότερες, οι περισσότερες απαντήσεις ήταν πως μπορούν να τιμωρηθούν ήδη με βάση την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία και επίσης κάποιες διοικητικέ δομές κρατών μελών απαιτούσαν περισσότερο χρόνο για εφέτηση, επίσης η πολυπλοκότητα του κανονισμού και βεβαίω η γνωστή αυτή καθυστέρηση στην εθνική νομοθετική διαδικασία. Άλλε Άλλες ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Περνάμε στο σημείο 8, στα ζώα λέει ο πρόεδρο. Ερωτήσει, Ζέμπερ, Λούκας και Έκουτ για τη, τα πειράματα που έχουν να κάνουν με ζώα. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα ερωτήματα Έκουτ, Λούκας και Ζέμπα. Η απάντησή μας θα ήταν ότι βάσει των συνεχιζομένων συζητήσεων μέσα στην ΕΚΑ και τις συζητήσεις μας με την ε, βιομηχανία και άλλους εμπλεκόμενους για το ΡΙΤΣ, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι ο αριθμός ζώων που υπολογιζόταν στην αρχή ότι θα χρησιμοποιούνται για να επιτυχθούν οι στόχοι του ΡΙΤΣ, ότι θα είναι πράγματι στην πράξη πολύ ψηλότερος. Αν τα ερωτήματα από τη δημοσίευση του καθηγητού Χάρτουγκ, η δική μας εντύπωση είναι ότι πολλές από τις επικρίσεις του κ. Χάρτουγκ δεν είναι τεκμηριωμένες. Εμείς συμφωνούμε με την ΕΚΑ όταν λέει στην ανακοίνωση τύπου της ότι η νέα αυτή μελέτη έχει υπερεκτιμήσει τον αντίκτυπο της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις δοκιμασίες σε ζώα κατά έξι φορές. Τα πραγματικά στοιχεία είναι μάλλον αυτά τα οποία είχαν δημοσιευθεί όταν είχε γίνει διαπραγμάτευση της νέας νομοθεσίας και αυτό λέει η δήλωση της ΕΚΑ. Τώρα είναι μια πολιτική, ένας πολιτικός συμβασμός μεταξύ μιας πληθώρας στόχων, καταρχήν προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος και δεύτερον την προώθηση εναλλακτικών μεθοδών δοκιμασίες. Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους έχει αναπτυχθεί ο κανονισμός του REACH ήταν ότι πολλές ουσίες είχαν παραχθεί και τεθεί σε εμπορία για πολλά χρόνια και έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες για τους ενδεχόμενου κινδύνους που θέτουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη να καλύψουμε αυτά τα κενά για να εξασφαλίσουμε ότι η βιομηχανία είναι σε θέση να εκτιμήσει τους κινδύνους και τους ενδεχόμενου κινδύνους και να εφαρμόσει την κατάλληλη διαχείριση κινδύνων και ενδεχομένων κινδύνων για να, να προστατεύσει τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η Κομισιόν πάντα ήταν σαφής ότι για να μπορέσουν να καλυφθούν αυτά τα κενά γνώσεων για τις χημικές ουσίες, το REACH θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη χρήση ζώων στα εργαστήρια, πειραματοζώων στα εργαστήρια τα επόμενα χρόνια, μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Αυτό ήταν γνωστό και έγινε δεκτό όταν συζητήθηκε το REACH από την αρχή της διαδικασίας αυτής. Για να μπορέσουμε όμως να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των δοκιμασιών σε ζώα, ο κανονισμός του ΡΙΤΣ περιλαμβάνει μια σειρά από ρήτρες για την προσαρμογή των αναγκών σε δοκιμασίες και να χρησιμοποιήσουμε τα τωρινά δεδομένα για εναλλακτικέ ε, μεθόδους δοκιμασίες. Τα τεστ σε σπονδυλωτά ζώα γίνονται μονάχα όταν δεν υπάρχει καμία άλλη ε, δυνατότητα και δεν θα επαναληφθούν τεστ τα οποία έχουν γίνει. Οι πληροφορίες αυτές λοιπόν θα διαμοιραστούν μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μέσω του συστήματος CF. Επίσης το παράτημα 11 περιλαμβάνει το πότε και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι ε, δοκιμασίες για να αντικαταστήσουν τις δοκιμασίες πειραματόζωα. Η Κομισιόν εμπλέκεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για να μειωθεί ο αριθμός των δοκιμασιών σε ζώα και να ε, εφαρμοστούν νέες διαδικασίες. Αυτό περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του GRC, τα ερευνητικά προγράμματα βάσει του προγράμματος πλαισίου έρευνας 7 και επίσης τις δραστηριότητες του ΟΣΑ στον τομέα αυτό. Τέλος θέλω να πω ότι η Κομισιόν υπέβαλε πέρσι μια πρόταση η οποία έχει σαν στόχο να εφαρμοστούν περαιτέρω οι διαδικασίες για τη μείωση και την αντικατάσταση των δοκιμασιών σε πειραματόζα για να μειωθούν τα βάσανα αυτών των ζώων. Η κυρία Λούκας. Ε, συμπληρωματικό ερώτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ήταν υπερβολική αυτή η εκτίμηση, αλλά ακόμα και αν ήταν, ο αρχικός αριθμός των, ε, των ζώων που είχαμε, ε, ε, υπολογιζόταν θα χρησιμοποιηθεί για το ρίτσι είναι ιδιαίτερα υψηλό. Και με, ανησυχούν, με ανησυχεί το γεγονό ότι δεν απαντήσετε και στι δύο ερωτήσει. Πρώτον, τι κάνετε για να επιταχύνετε ε, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών μοντέλων, συμπεριλαμβάνοντα μεθοδολογίες ε, όπως ε, για παράδειγμα ε, τοξική ανάλυση και δεύτερον τι κάνετε με την έκθεση 2007 της, Ακαδημαϊκής, της Ακαδημίας Επιστημόνων για την τοξικότητα. Γιατί μεγάλο μέρος αυτής της έκθεσης αφορά το θέμα της επαλήθευσης. Άρα συμπληρωματική ερώτηση είναι εξή. Τι κάνει η Επιτροπή για να διερευνήσει νέε προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση, την αποτελεσματικότητα των μεθόδων, όπου δεν είναι σωστή δηλαδή, όπου δεν είναι κατάλληλη η συμβατική επαλήθευση. Και δεύτερον, ανθρώπινα στοιχεία που προέρχονται από κλινικέ δοκιμέ φαρμάκων θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και πώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδό για να αξιολογήσουμε τι επιδόσει των, αποτελεσματικότητα των φυσικολογικών μελετών και στα ζώα και εκτό των ζώων. Γιατί ε, ο χρυσό κανόνα είναι ακόμα τα πειράματα σε ζώα. Ε, και όμω είναι σαφέ ότι ε, ε, τα εμπειρικά δεδομένα για την, για την έκθεση των ανθρώπων ε, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά. Και επειδή αυτά συλλέγονται κάτω από πολύ αυστηρέ συνθήκε και ήδη συλλέγονται, γιατί δεν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο ω τον ε, βασικό κανόνα. Θέλω λοιπόν να απαντήσετε στι δύο πρώτε ερωτήσει σύν σε αυτέ τι δύο συμπληρωματικέ. Ε, Πρόεδρε, έχω την εντύπωση, είχα την εντύπωση ότι είχαμε απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν, αλλά μάλλον κάνουμε λάθος. Με την έννοια ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου που έθεσαν τα ερωτήματα. Τι να κάνω, να επαναλάβω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαμε. Όταν εγκρίθηκε το ΡΙΤΣ, όλοι γνωρίζαμε τι ακριβώς θα γινόταν, αλλά μετά από το 14 χρονικό διάστημα, ότι θα είχαμε τη μείωση. Οι λόγοι είναι αυτοί που σας ανέπτυξα. Ότι υπάρχουν κενά στη γνώση μας. Για να συμπληρώσουμε αυτά τα κενά, αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε τα πειράματα στα ζώα. Και εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή βασικά. Τώρα, συμφωνούμε απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο οργανισμός. Όσον αφορά αυτή την αντίδραση στο άρθρο, είναι πολύπλοκες αυτές οι σχετήσεις με τις οποίες δεν συμφωνούν οι εμπειρογνώμονες. όσον αφορά ε, το πού βρήκαμε αυτούς τους αριθμούς. Τώρα, ε, ε, από μερικές Αμερικής. Να σας διαβάσω το εξή. Ιδιαίτερα το παράρτημα 11 του ΡΙΤΣ αναφέρεται στην άμεση εφαρμογή εναλλακτικών μεθοδολογιών όπως αυτές που αναφέρονται στην έκθεση του Εθνικού Φορέα της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών εφόσον βεβαίω οι μεθοδολογίε ε, απαντούν στα βασικά ερωτήματα εντοπισμού δηλαδή του κινδύνου που προέρχεται από τι χημικέ αυτέ ουσίε. Δηλαδή δεν πέρασε παρατήρητο στοιχείο αυτό. Είναι βασικό στοιχείο του προβληματισμού μα και αναφέρεται στο παράδειγμα 11. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Αντίκτυπος του Ριτς στο περιβάλλον και την υγεία. Ο κύριος Ζέμπερ έχει παρόλα αυτά ε, μία ακόμα ερώτηση για τα ζώα. Ναι, υπάρχει αυτό το άρθρο του καθηγητή Χαρτινού στο Nature που προξένησε διάφορες αντιδράσεις. Θέλω να γνωρίζω από την Κομισιόν συγκεκριμένα πόσα χρήματα έχετε αφιερώσει για να προωθηθούν οι εναλλακτικέ μέθοδοι έρευνας τα τελευταία πέντε έτη. Πόσα λεφτά έχουν πάει για τις εναλλακτικέ μεθόδους ε, δοκιμών. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω τα νούμερα μαζί μου. Θα σας τα στείλουμε αργότερα κάποια στιγμή αυτό ψάξουμε. Θα τα λάβουμε αργότερα λοιπόν κύριε Ζέιμπερ. Παίρναμε στο επόμενο σημείο επιδράσεις του ΡΙΤ στο επιβάλλον και την υγεία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έχετε να μας πείτε κάτι, να απαντήσετε κάτι εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και τις επιχειρήσεις και μετά ο συνάδελφος θα μπορούσε να συμπληρώσει για τα λοιπά. Ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να διακρίνουμε δύο επίπεδα. Έχουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας καθεαυτή και μετά εάν υπάρχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους ανταγωνιστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του REACH. για να ξεκινήσω από το δεύτερο, δεν έχει εισαχθεί καμία υποχρέωση στο REACH μόνο για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και που δεν θα επηρεάζουν τους ε, παραγωγούς των ίδιων χημικών ουσιών εκτός ένωσης ε, που κάνουν εξαγωγές. Οπότε έχουμε δημιουργήσει ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για να μην υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος ανάλογα με το πού παράγεται το προϊόν. Για την ανταγωνιστικότητα της ε, βιομηχανίας χημικών είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να κάνω σοβαρό σχόλιο γιατί ακόμα προετοιμάζονται οι φάκελοι για την ε, καταγραφή απέχει ακόμα ένα χρόνο η προθεσμία. Δεν υπάρχει λοιπόν άμεσο αντίκτυπο. Μόνο εκ των υστέρων θα μπορέσουμε να πούμε ποιο είναι το πραγματικό κόστο και η επίδραση. Αλλά οπωσδήποτε ε, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι πως το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης ε, και της γενικότερης πτώσης είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του ΡΙΤΣ, οπότε πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί να μην επιβαρύνουμε τη βιομηχανία με ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. Και απ' την άλλη μας απασχολεί γενικά η ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας και εκεί πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ η ομάδα υψηλού επίπεδου περί ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας που ολοκλήρωσε πέρσι τις εργασίες της και θα δούμε και θα ακολουθήσουμε τις ε, συστάσεις της. Τώρα για τις ε, επιπτώσεις στη φύση θα δώσω τον λόγο συνάδελφο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έκανα ήδη μία ανοίξη όταν απάντησα στον κύριο Ζέμπερ ότι το παρακολουθούμε ενεργά. Έχουμε κάνει μία βασική μελέτη για, το που, για να έχουμε μία φετηρία δηλαδή και μετά μπορούμε να συγκρίνουμε το, τις εξελίξεις τις μελλοντικέ θα έχουμε μια δεύτερη μελέτη που προβλέπεται για το 2012 οπότε έχουμε ένα ενεργό μέσο για να δούμε ποια επίδραση θα έχει το ΡΙΤΣ ε, στην υγεία και τη φύση. Yeah. Ωραία. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν. Έχουμε το ερώτημα του κυρίου Περίγιο τις επιπτώσεις σε άλλα πεδία νομοθεσίας και η κυρία Λεπάζ και ο κύριος Σλίτορ έχουν θέσει ερωτήματα για τα νάνο Αν μπορώ να ξεκινήσω με τη σχέση με άλλα νομοθετήματα και να περάσουμε τα στα νανοηλικά, το ριτς δεν είναι η απαρχή της χημικής νομοθεσίας, αλλά αντικαθιστά 40 νομοθετήματα τα οποία είναι ενισχύ ήδη. Επομένως, το REACH δεν αντιμετώπισε όλες τις χρήσεις χημικών ουσιών, όπως τα φαρμακευτικά σκευάσματα ή στα τρόφιμα, αλλά με την επιφύλαξη της νομοθεσίας στο περιβάλλον, έχει αφήσει αυτά τα θέματα απ' έξω. Υπάρχουν ορισμένα νομοθετήματα λοιπόν, όπως πραγματικά για τα καλλιντικά, η οδηγία για τα καλλιντικά ο κανονισμός για τα καλλιντικά ή για τις οικολογικές ετικέτες που δεν αντικαθιστώνται από το Ο νομοθέτης έχει κάνει μια σαφή οριοθέτηση του τι καλύπτει το ΡΙΤΣ και τι δεν καλύπτει. Και συγχρόνως η διαδικασία του ΡΙΤΣ θα καθορίσει, θα δημιουργήσει μια μεγάλη βάση δεδομένων για τις χημικές ουσίες και τις ιδιότητές τους, κάτι το οποίο θα βοηθήσει την εφαρμογή των άλλων νομοθετημάτων και την επίτευξη των στόχων τους. Έτσι αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους καταναλωτές στον τομέα των καλλιντικών παραγωγής χάρη και για την ε, ετικετοθεσία που οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια στον χώρο εργασίας και για άλλη περιβαλλοντική νομοθεσία θα είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσω ότι η Κομισιόν αντιμετωπίζει με μεγάλη προσοχή τη σχέση αυτού του νομοθετήματος με τους άλλους τομείς νομοθεσίας ιδίω όταν προχωρούμε σε αναθεώρηση ή τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις ή νομική ασάφεια η οποία δημιουργείται με την εφαρμογή του συστήματος REACH. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την εφαρμοσιμότητα στα να νανοηλικά της αρχής ότι αν δεν υπάρχουν στοιχεία δεν τίθενται σε εμπορία. Πρέπει να σας πω ότι αυτό εφαρμόζεται σε ουσίες, είτε είναι μεμονωμένες είτε είναι σε μείγματα, είτε σε άλλες μορφές. Εφαρμόζεται λοιπόν αυτό και στα νανοηλικά. Δηλαδή οι φάκελοι εγγραφής αφορούν τα νανοηλικά που μπορούν να είναι αυτόνομα υλικά ή μέσα σε άλλε ουσίε και θα πρέπει εκεί να περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και νανοπληροφορίες για αυτά τα υλικά. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, προστασία του περιβάλλοντος, ελεύθερη αντα... κυκλοφορία, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Πολλά νανοηλικά παράγονται με ιδιαίτερα ε, καινοτόμες τεχνικές που βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος, μπορούν να δώσουν πολλά πλεονεκτήματα για προϊόντα που προορίζονται για του καταναλωτέ και επίση μπορούν να βελτιώσουν την προστασία του περιβάλλοντο. Υπάρχουν όμω και ορισμένε ανησυχίε για την ασφάλεια αυτών των ανοηλικών που θα πρέπει να τύχουν τη σωστή διαχείριση για να υπάρξει η ανάπτυξη αυτή τη τεχνολογία με τρόπο βιώσιμο. Στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου τη 24η Απριλίου ζητάτε από την Κομισιόν να αναθεωρήσει και να εξετάσει όλη την νομοθεσία σε σχέση με τα νανοηλικά για να εξασφαλίσει την ασφάλεια σε όλες τις εφαρμογές των νανοηλικών σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μέσα στον κύκλο ζωή αυτών των ανοηλικών. Η Κομισιόν έχει σαν στόχο να αναθεωρήσει και να εξετάσει όλη αυτή την νομοθεσία και την εφαρμογή τη και να δώσει μια έκθεση για όλα αυτά το 2011 όταν θα προταθούν οι απαραίτητο οι αλλαγέ στα νομοθετήματα αυτά. Η Κομισιόν φυσικά αποδίδει μεγάλη σημασία σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία απασχόλησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άλλα ερωτήματα, ο Καρλ Σλούτερ. Ναι, θα είμαι σύντομος, λέει ο Καρλ Σλούτερ. Λέτε ότι το ριζ καλύπτει ένα συγκεκριμένο πεδίο. Έχετε <coughs> ασχοληθεί με το εύρος των τοξικολογικών δοκιμασιών. Αν καλύπτουν ορισμένες ιδιότητες των νανοηλικών. Μήπως μπορείτε να επανέλθετε στο θέμα αυτό. Και επίσης, αν είναι δύο χρόνια, 24 Απριλίου 2011 είναι Κυριακή. Επομένως τη Δευτέρα θα πρέπει να έχετε περατώσει αυτή τη διαδικασία. Την επόμενη Δευτέρα δηλαδή. Κύριε Μπόσετ. Εμένα το, η ατζέντα μου σταματάει πριν από τον Απρίλιο του 2011. Εμείς ε, συμμετέχουμε ιδιαίτερα ενεργά στο θέμα αυτό και στην εξέλιξη των ε, συζητήσεων μέσα στον ΩΣΑ. Όταν καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, δεν θα βραδύνουμε να πληροφορήσουμε τον αξιότιμο κύριο Βουλευτή για τα πορίσματα των συζητήσεων αυτών. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Έχει κλείσει λοιπόν ο γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων για το ΡΙΤΣ που είναι στρατηγικός ακρογωνιαίος λήθος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλες αυτές οι ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο περιβάλλον και στην αγορά θα πρέπει να καταγραφούν και να τύχουν ελέγχου. Ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει αυτός ο μηχανισμός για την καταγραφή αυτή με επιτυχίες αλλά και με προβλήματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά γιατί είναι τεράστια η πολυμορφία και η πολυπικιλία αυτών των ουσιών Ακούσατε τα ερωτήματα όλων των συναδέλφων. Η Επιτροπή μας φυσικά θα παρακολουθήσει από πολύ κοντά όλα αυτά τα θέματα και στο μέλλον και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Διευθυντή του Φορέα για τις Χημικές Ουσίες το Νοέμβριο. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε και πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Ευχαριστώ λοιπόν τους εκπροσώπους της Κομισιόν που ήλθαν εδώ και απήντησαν τα ερωτήματα αυτά. Ελπίζουμε ότι σε ένα μεταγενέστερο επίπεδο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την επωφελή εργασία. Και ερχόμαστε τώρα αγαπητοί συνάδελφοι στο σημείο, στο επόμενο σημείο, πάση περιπτώσει μέση διάταξη, το σημείο υπάρχει μόνο 8. Σχέδιο ενός μέτρου επιτροπολογίας βάσει της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα πλαίσια της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής και πρόκειται για τον κατάλογο των τομέων και επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως λέγεται, δηλαδή μετακίνησης επιχειρήσεων. Είναι η προβληματική αυτή η οποία αναφέρεται λοιπόν ως διαρροή άνθρακος. Και τώρα στο θέμα αυτό έχουμε την Ιβόν Σβίγγενμπεργκ και ο Χάνς Μπέργμαν και ο Ντάνιελ Μέντος από την Κομισιόν από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και θα πρότεινα να λάβει η Κομισιόν τον λόγο πρώτα να μας παρουσιάσει την κατάσταση των πραγμάτων και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ευρύτερη συζήτηση. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει από την πλευρά της Κομισιόν. Ο Ντέμιαν Μέντος. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Η Κομισιόν με μεγάλη χαρά θέλει να παρουσιάσει αυτό το οποίο πιστεύω είναι το πρώτο νομοθετικό μέτρο το οποίο εφαρμόζει το πακέτο ενέργειας και κλιματικών θεμάτων που ενεκρίθη πέρσι. Αυτός ο κατάλογος των βιομηχανιών, οι οποίες θεωρείται ότι εκτίθενται σε, μέσα σε εισαγωγικά διαρροή άνθρακος, ήταν ένα κομβικό θέμα στο διαπραγματεύσεων που, στο που οδήγησαν σε συμφωνία πέρσι με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να θεσπίσουν μια καταληκτική προθεσμία 31 Δεκεμβρίου του 2009 για να υπάρξει αυτός ο κατάλογος. Για να το κάνουμε αυτό το πράγμα, εμείς εργαστήκαμε ιδιαίτερα εντατικά, με μεγάλη στενότητα χρόνου. Υπήρξαν οι προτάσει των ε, κρατών μελών προ την Κομισιόν που ήρθαν εγκαίρω και η παρακολούθηση από το Κοινοβούλιο επίση έχει γίνει έγκυρα, έγκαιρα ώστε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτό το κατάλογο στι 23 Δεκεμβρίου που είναι η τελευταία εργάσιμη ημερομηνία του 2009. Λόγω όμω του χρονοδιαγράμματος που απαιτείται για αυτό το θέμα πριν από τη διάσκεψη της Κοπενχάγης και πριν δοθεί πλήρης πληροφόρηση για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, ο κατάλογος αυτός μπορεί να αναθεωρηθεί μετά από τα αποτελέσματα της Κοπενχάγης. Και είμαστε έτοιμοι για ένα σενάριο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει μόνη της στην μονομερή της δέσμευση για μείωση 20% για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου μας ε, ενθαρρύνει η προσπάθεια που κατεβάλλεται από άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά εάν δεν υπάρξει καμία συνεργασία από άλλες χώρες, ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να ισχύει μέχρι το 2014 και οι άλλες, άλλοι τομείς μπορούν να προσθεθούν βάσει επιτροπολογίας, αλλά κανονικά δεν μπορούν να, να αφαιρεθούν από τον κατάλογο. Ένας νέος κατάλογος θα ισχύει για το χρονικό διάστημα 2015-2019. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του καταλόγου αναφέρονται 164 βιομηχανικοί τομεί και υποτομεί, επιμέρου τομεί, οι οποίοι βάσει των λεπτομερών κριτηρίων στην οδηγία θεωρούνται ότι έχουν εκτεθεί σε διαρροή άνθρακα. Αυτή δεν είναι διαδικασία όπου η Κομισιόν είχε ιδιαίτερη διακριτική ευχέρεια, γιατί τα κριτήρια έχουν θεσπιστεί από το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως αποφασίστηκε πέρσι. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να εμπλέξουμε όλους τους εμπλεκόμενους για την ανάπτυξη αυτού του καταλόγου και στην ιστοσελίδα μας και επίσης στην ε, ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο έχουμε πλήρη τεκμηρίωση και δελτία ε, κτλ. Και έχουμε επομένω και ανακοίνωση που Μπορούμε θαυμάσια λοιπόν να εξηγήσουμε πώς καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει. Τέλος θα ήθελα να πω για τον κατάλογο αυτό ότι πρέπει να τονίσω ότι αυτή η, ο κατάλογος αυτός αντανακλά την καλύτερη, το, το βέλτιστο επίπεδο γνώσεων που έχει καταφέρει να συλλέξει η Κομισιόν μέχρι στιγμή σε συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Καταλήξαμε και σε μια αιτιολογική σκέψη που λέει ότι μπορούν και θα προσθεθούν τομείς βιομηχανικοί σε αυτόν τον κατάλογο αν υπάρχουν τεκμήρια που να το στηρίζουν. Η Κομισιόν πάντως έχει αναλύσει εξονυχιστικά τον κατάλογο αυτό των 164 τομέων και επιμέρους τομέων που είναι αυτοί που ε, αντιστοιχούν στα κριτήρια της οδηγίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να ε, χαιρετήσω και την ομάδα των ε, εμπλεκομένων που εκπροσωπείται εδώ μέσω της κυρίας Κέλλη. Θα ήθελα λοιπόν εξ ονόματος της Επιτροπής μας να σας καλωσορίσω στην συνεδρίασή μας σήμερα. Και έχουμε τώρα τον Πέτερ Λίζε, ο οποίος θα λάβει το λόγο καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που βάλατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ε, συζητήσεις και κριτικές παρατηρήσεις από δύο πλευρές και από τη βιομηχανία και από τις ε, ΜΚΟ. Με βάση αυτά τα οποία μέχρι στιγμής γνωρίζουμε και διαβάσαμε και την ε, αντίδραση των διαφόρων ενδιαφερομένων είναι λογική η απόφαση που έλαβε η Κομισιόν, η πρόταση δηλαδή που κάνει. Θεωρώ πως η Κομισιόν τήρησε την εντολή της που τις έδωσαν δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλοι μαζί από κοινού και εδώ απευθύνω έκκληση της ε, ΜΚΟ να μην ε, κακολογούμε την απόφαση της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλιματικό πακέτο. Έχουμε πει πως θα μείνουμε στο 20% αν είμαστε μόνοι μας και 30% αν υπάρξει συμφωνία. Η νέα Ιαπωνική κυβέρνηση, δόξα τω Θεώ, γιατί ήταν και αναγκαίο, αύξησε το στόχο της στο 25% αλλά δεν έχει κάνει καμία προσφορά να προχωρήσει παραπάνω εάν είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Στις ΔΕΗ, όπως ξέρουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει αυτός ο νόμος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ε, που προβλέπει μείωση κατά 10% ακόμα και αυτό είναι δύσκολο. Οπότε αυτό το 20% και η διαθεσιμότητά μας να πάμε και στο 30% δεν είναι τέλειο και δεν είναι το τέλος στο οριστικό της συζήτηση, αλλά είναι πολύ φιλόδοξο με βάση τα οποία έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή και μέρος αυτού του συμβασμού ήταν πως θα πρέπει να βοηθεί αυτή η διαρροή μετακίνηση δηλαδή επιχειρήσεων και θα πρέπει άρα κάποιοι τομείς να εξαιρεθούν από τη δημοπρασία, όχι από το στόχο. Και πρέπει να το πούμε αυτό και προς τα έξω όταν βλέπουμε την συνολική πρόταση της ε, Κομισιόν, γιατί δεν πρέπει να επιβαθμίσουμε και την δική μας την διαπραγματευτική θέση, γιατί απομακρυνόμαστε έτσι από το στόχο μας. Δεν είναι διαφορετικός ο στόχος, είναι θέμα μεθόδου απλά. Και βεβαίω όλοι γνωρίζουμε πως χρειαζόμαστε λεφτά ε, για την Κομεχάγη, γι' αυτό πρέπει να έχουμε και δημοπρασία, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα βεβαίως των εκπομπών στο εμπόριο εκπομπών πρέπει να δημοπρατηθεί είτε γιατί θα ξεκινήσουμε άμεσα όσον αφορά τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από το 2013 είτε για το ότι οι διάφοροι παραγωγικοί τομείς θα ακολουθήσουν επίσης το 50% των εκπομπών δεν καλύπτονται καν από το σύστημα εμπορίας ε, το 50% των εκπομπών της Ευρώπης και θα πρέπει και αυτοί οι τομείς ε, να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της Κοπενχάγης. Οπότε θεωρώ πως είναι λογικός ο συμβασμός. Έχω όμως και κάποιες ερωτήσεις για την Κομισιόν. Σε ένα έγγραφο ενημέρωση των NGO διάβασα πως, των ΜΚΟ πως εάν δεν είναι επιτυχής η κατάληξη της Κοπενχάγης, κάτι το οποίο είναι πιθανό. Αλλά εάν καταφέρουμε παρόλα αυτά να περάσουμε και στις τρίτες χώρες την δημοπρασία, ακόμα και τότε δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάποια αναθεώρηση. Ο κύριος Μέντος μας είπε πως δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο κατά την άποψη Κομισιόν. Θα ήθελα όμως να ακούσω την άποψη της Κομισιόν. Εάν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα στην Κοπεχάγη που θα οδηγήσει σε δημοπρασία σε αυτές τις ε, βιομηχανίες, θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψή μα, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δεν υπάρχει καν ε, στην ημερήσια διάταξη η δημοπράτηση, αλλά θα υπάρξει μια προσαρμογή πρώτον. Και δεύτερον, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τομεί ε, στην βιομηχανία οι οποίοι με ένα στόχο 20% ε, δεν καλύπτονται από την διαρροή. Οπότε, εάν το οξύνουμε κάπως το πράγμα και συμφωνήσουμε ε, βεβαίως, αλλά δεν είναι συγκρίσιμη η βάρεση της βιομηχανίας. Πώς θα ρυθμιστεί το ζήτημα, πώς θα προχωρήσουμε σε 30% μείωση χωρίς ε, δημοπράτηση. Υπάρχουν τομεί που κινδυνεύουν να φύγουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ είναι οι δύο ερωτήσει μου. Η τρίτη μου ερώτηση για την Κομισιόν. 77% των εκπομπών καλύπτονται από την ειδική αυτή μεταχείριση. Δεν είναι όμως 77% των επιχειρήσεων. Δηλαδή αν δούμε το κλάδο του τσιμέντου παραδείγματος χάρη εξαιρείται γιατί έχει τόσο μεγάλο ποσοστό εκπομπών όσον αφορά την υπεραξία του. Το, το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες επιχειρήσεις, αλλά ήθελα να ξέρω πόσο ποσοστό των επιχειρήσεων εξαιρείται και ποιοι κλάδοι είναι υποψιολογικές συνθήκες ε, στην ε, δημοπράτηση αυτή, δηλαδή ποιοι, ποιοι τομείς ε, θα συμπεριληφθούν κανονικά υποκανονικές συνθήκες. Ευχαριστώ θα ακούσουμε τρεις-τρεις ερωτήσεις. Να καλωσορίσω λοιπόν την Evelyn Doyle, η οποία ήταν η συγγήτρια για το ζήτημα του συστήματος εμπορίας εκπομπών, οπότε βεβαίως την απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και εφόσον τελείωσε και το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία είναι ελεύθερη να ασχοληθεί και με άλλα ζητήματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ε, κατόπιν να ακούσουμε τον Μητόριο Πρόντι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι διαφωνώ με αυτό το έγγραφο γιατί πιστεύω ότι στην Κοπενχάγη πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα εξέβρισης συνολικής συνένεσης. Οτιδήποτε λιγότερο δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτα. Τώρα, επομένως θα πρέπει να δούμε ευθύ εξ αρχή. Τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση διαρροή άνθρακα. Αυτό αποτελεί αποδυνάμωση, αν θέλετε, ε, αυτής, ε, ε, της ανάγκης που υπάρχει να, για συνολική λύση. Στην περίπτωση βέβαια αυτή τη τελευταία, τη συνολικής λύσης, συμπεριλαμβάνουμε και τη διαρροή του άνθρακα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα της συνολικής λύσης και νομίζω ότι για την Κοπεχάγη λείπουν, ορισμένα βασικά, λείπουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα ρήτρα ισοτιμίας, ακριβώς διότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν επαρκής εγγυήσεις για το ότι το δικαίωμά τους στην ανάπτυξη θα γίνει σεβαστό. Δεύτερον, πιστεύω ότι και ήδη ε, το έχω αναφέρει και γραπτά στον πρόεδρο της Επιτροπής, στον κύριο Μπαρόζο. Πιστεύω λοιπόν ότι ότι αυτός ο έλεγχος των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου και αυτό το σύστημα είναι ε, ιδιαίτερα ε, κατατμημένο. Εμείς χρειαζόμαστε ένα πιο γενικό και πιο απλό σύστημα. Δηλαδή κάθε χρήση ε, ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να υπόκειται σε, αυτό, σε αυτούς τους περιορισμούς. Δεν τίθεται ζήτημα λοιπόν εξαιρέσεων. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το θέμα της ισοτιμίας και της γενικής κλιματικής δικαιοσύνης, αν θέλετε. Βεβαίως ε, ε, θα πρέπει ε, να πετύχουμε ένα βιώσιμο σύστημα και όσον αφορά τις εκπομπές κατά κεφαλήν από τους 5 τόνους ισοδύναμων εκπομπών άνθρακα θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα τόνο μονοξιδίου του άνθρακο ανά άτομο και ανά έτος. Εάν αυτό θεωρέσουμε ότι είναι εφικτό επίπεδο, τότε σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε άτομο, ακριβώς για τους, λόγου κλιματική λόγους κλιματικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να αποδοθεί το ίδιο δικαίωμα χρήση των φυσικών πόρων. Άρα και της ατμόσφαιρας. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς θα πρέπει να δώσουμε δωρεάν, αν θέλετε, άδεια εκπομπών ε, δύο τόνων μονοξιδίου του άνθρακος ανά άτομο ε, ανά έτος, ε, δύο τόνους, άρα λοιπόν και οξυδιού του άνθρακος, άρα λοιπόν χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την Αφρική που βρίσκεται πολύ κάτω από, τον, από το ποσό αυτό, άρα θα πρέπει να θέσουμε στην αγορά γύρω στους 0,8 τόνους ανά άτομο, ανά έτος. Άρα λοιπόν παίρνοντας άμεση συνεισφορά που θα είναι ουσιώδους σημασίας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιματική αλλαγή που αυτή τη στιγμή ισοδυναμεί με 15 δις ευρώ το χρόνο. Άρα λοιπόν βλέπετε το πώς ε, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε καν να έχουμε την ελπίδα ότι θα έχουμε αυτή τη συνολική συμφωνία στην Κοπεχάγη. Και ε, αυτό θέλω να σκεφτεί η ομάδα και η Επιτροπή. Γιατί χωρί αυτέ τι ρήτρε ισοτιμία, η συμφωνία στην Κοπεχάγη δεν θα μα χρησιμεύσει τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι η Κομισιόν διατυπώνει το στόχο Εάν δεν, υπάρξουν, δεν υπάρξει συμφωνία με τις άλλες χώρες που είναι μεγάλοι ρηπαντές με διοξίδιο του άνθρακος, θα υπάρξει το θέμα της μετακίνησης των επιχειρήσεων προς χώρες όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Η λεγόμενη διαρροή άνθρακος. Βέβαια, όταν συζητήθηκαν αυτά τα θέματα, ενέργεια και κλιματική αλλαγή μαζί, ήταν να εξασφαλίσουμε παγκόσμια τις ίδιες προδιαγραφές και όχι να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα έφτανε στα όρια αυτών που είχαν συμφωνηθεί με το κλιματικό πακέτο και θα αναγκαζόμασταν να επανέλθουμε στα προηγούμενα επίπεδα των ε, ε δυνατοτήτων εκπομπή μέχρι το 100% που οδήγησε σε επικρίσει για το σύστημα εμπορία εκπομπών. Τα ερώτηματά μου τώρα είναι τα εξή. Μα είπαν ότι σε ορισμένε περιπτώσει δεν υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν μονάχα ιδιωτικές μελέτες που έχουν γίνει. Τι κάναμε για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αυτά τα στοιχεία. Δεν ήταν σαφές από αυτά που είπε η Κομισιόν το πώς θα προχωρήσουν στους τομείς αυτούς όπου ελείπουν τα απαραίτητα δεδομένα. Και επίσης λέει η Κομισιόν ότι ορισμένοι βιομηχανικοί τομείς θα εξεταστούν μονάχα το 2010. Ποια είναι η πρόγνωση, ποιες είναι οι προβλέψεις για τις προτάσεις από τις οι οποίες θα προκύψουν από αυτή την ε, εξέταση, τι ποσοστό από αυτούς τους τομείς θα συμπεριληφθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και ποιοι τομείς θα πάρουν 100% ε, άδειες εκπομπής. Υπάρχει εδώ μια σαφής διαδικασία για να καταλήξουμε σε την επιβολή υψηλών προδιαγραφών για όλους και όχι μια αποδυνάμωση των κριτηρίων αυτών και μια επαναφορά δυσκολιών που θα είχαμε στις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες όταν τους δούμε να πάρουν κάποια μέτρα και μετά μπορούν να μας υποδείξουν τις δικές μας δυσκολίες σε τομείς όπου εμείς θεωρούσαμε ότι εκεί θα μπορούσε να αναλυφθεί υψηλό επίπεδο ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την Κομισιόν να απαντήσει, κύριε Στρίνμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ήδη ε, ακούσατε ε, την εισαγωγή για το θέμα αυτό από τον αναπληρωματή μας. Ευχαριστώ λοιπόν τα μέλη του Κοινοβουλίου για τις ερωτήσεις σας. Ίσως λοιπόν θα, θα μπορούσαμε να, τι δούμε κάπως με την ε, σειρά που ετέθησαν. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο κατάλογος είναι ο πρώτος κατάλογος κατά κάποιο τρόπο προβλέπεται στην οδηγία για αναθεώρηση, η οποία προβλέπεται στην οδηγία για αναθεώρηση, που θα λάβει η χώρα με τρει διαφορετικού τρόπου. Ο πιο σημαντικό, στον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Γλίζε, είναι το γεγονό ότι μετά την Καποχάγη η Επιτροπή ε, έχει λάβει την εντολή να αξιολογήσει το αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων και να δει κατά πόσον υπάρχει συγκεκριμένο αντίκτυπο στην προσέγγιση που είχαμε μέχρι στιγμή. Άρα λοιπόν, αυτό θα το πράξει η Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτου. Θα υποβάλει δηλαδή έκθεση και θα δούμε κατά πόσον η έκθεση μέχρι στιγμή ε, ευσταθεί ή πρέπει να ε, προσαρμοστεί. Και σίγουρα αν υπάρξει καλή συμφωνία από την Κοπενχάγη θα εξετάσουμε πολύ μεγάλη προσοχή το κατά πόσον υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό κίνδυνο για διαρροή άνθρακα σε όλου αυτού του τομεί ή κατά πόσον έχει μειωθεί. Και αυτό βεβαίω θα εξεταστεί, για παράδειγμα, μέσω ε, των στοιχείων έκθεση του εμπορίου. και και αν δηλαδή και οι τρίτε χώρε έχουν λάβει σημαντικά μέτρα και κατά πόσο ε, και αυτά βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο προ του στόχου. Στα δεδομένα τα εμπορικά θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε τι χώρε αυτέ ε, και μπορεί να έχουμε και ε, τομεί κάτω από 30% του κριτηρίου για την έκθεση. Άρα θα του αφαιρέσουμε από τον κατάλογο. Τέλο πάντων, προβλέπεται η αξιολόγηση Κοπεχάγη. Δεν έχω δει ακόμα το έγγραφο που στο οποίο αναφερθήκατε. Πάντω σίγουρα είναι πιθανό να το προσαρμόσουμε. Επίσης, αν δεν είναι ιδεώδε το αποτέλεσμα, θα δούμε και τι ανισότητε και, και την άνηση κατανομή του βάρου και αυτό προβλέπεται, ε, προβλέφθηκε στο πακέτο διαπραγματεύσεων του περασμένου έτου. Γιατί ε, αυτό το επίπεδο 100% για τις ε, ε δωρεάν ε, άδειε ε, και τις συγκριτικές μελέτες εξακολουθεί να υπάρχει. Θα δούμε όμως κατά, κατά πόσο απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα ή άλλα μέτρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ανοιχτά ζητήματα που θα εξεταστούμε μετά την Κοπεχάγη. Αναφερθήκατε στο γεγονό ότι 77% των εκπομπών καλύπτονται. Ποιο ποσοστό των εγκαταστάσεων, σα το χρωστάω αυτό το αριθμητικό στοιχείο. Θα πρέπει να δούμε τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται ε, στη, σε αυτό το ημερολόγιο το ανεξάρτητο των συναλλαγών τη Επιτροπής αλλά γύρω στο 50% ή κάτω από το 50%. Αυτέ είναι οι χοντρικές μα εκτιμήσει. Δεν είναι κάτι πάντω που το έχουμε ελέγξει λεπτομερίες του. Ε, οι κλάδοι που θα εξακολουθούν να υπόκειται το σύστημα δημοπράτησης είναι πολλοί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, ε, ότι δεν θα τεθούν εκτός συστήματος αυτοί που εκπέμπουν σε μεγάλο βαθμό. Ε, είχαμε συζητήσεις με πολλούς τομείς ή υποτομείς που αυτή τη στιγμή δεν είναι στον κατάλογο και ε, θα προτείνουμε τη συμπερίληψη και αυτών στον κατάλογο. Ε, υποτομέας ε, κεραμικών, ε, πλακάκια και τούβλα. Το ξέρετε το τομέα αυτό, θα τον απεναξιολογήσουμε βάσει των δεδομένων που θα μας δώσουν στους επόμενους μήνες. Ε, να άλλη μια αναθεώρηση στον κατάλογο, δηλαδή προσθήκη τομέων σε αιτήσια βάση και προφανώς θα εξετάσει οποιοδήποτε τομέα η Επιτροπή με πρωτοβουλία της Επιτροπής με πρωτοβουλία των κρατών μελών και θα προσθέσουμε όλους αυτούς ε, στον κατάλογο, εάν βεβαίω υπάρχει απόδειξη ε, ότι πληρούν τα κριτήρια. Σε αιτήσια βάση δεν προβλέπεται η αφαίρεση τομέων από τον κατάλογο. Καταρχήν ο κατάλογο ισχύει για πέντε χρόνια, με δύο εξαιρέσει. Ετήσιε προσθήκε ή πλήρη αναθεώρηση μετά την Κοπενχάγη. Που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, διαγραφή από τον κατάλογο ορισμένων. Τώρα, αυτά που ο κύριο Πρόντι για τις ισότιμες διατάξεις ε, που απαιτούνται για μια καλή συμφωνία στην Κοπεχάγη. Σημειώσαμε τις παρατηρήσεις του και πράγματι αυτό το στοιχείο ε, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή και στην Μπαγκόκ στις διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος που γίνονται εκεί αυτή τη στιγμή. Σημειώσαμε λοιπόν όλα αυτά που είπατε και θα δούμε ε, πού θα μας οδηγήσουν οι διαπραγματεύσεις. Βεβαίως είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο κατάλογος διαρροής άνθρακα πρότεινε η Επιτροπή το Σεπτέμβριο στηρίζεται ε, στο στόχο 20% ως γενικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, ε, μετά την Κοπενχάγη προκύψει να έχει υψηλότερο στόχο, βεβαίω θα προσαρμοστούμε. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τι δεσμεύσει των τρίτων χωρών. Στη συνέχεια είχαμε μία ερώτηση σε σχέση με τα στοιχεία και τι θα κάνουμε για να παίρνουμε καλύτερα δεδομένα. Εδώ στην ουσία μιλάμε για τους τομείς που είπαν ότι και αυτοί θα πρέπει να έχουν προσθεθεί στον κατάλογο θέλουμε να συνεργαστούμε με την βιομηχανία αλλά και με τα κράτη-μέλη για να έχουμε καλύτερα δεδομένα και θα δούμε κατά πόσον μπορούμε σε συνολική βάση να έχουμε καλύτερα δεδομένα και καλύτερα στοιχεία. Θα επεξεργαστούμε αυτή την πιθανότητα και τη δυνατότητα και βεβαίω ε, θα έχουμε και νέα στατιστικά στοιχεία. Έχουμε αυτή τη στιγμή ε, χρήση νέα ονοματολογία στα πλαίσια ε, μιας εξέλιξης Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να τονίσω το εξή κάτι ε, το οποίο, ε, για το οποίο πρέπει να διαλυθεί κάθε παρεξήγηση. Όταν μιλάμε για τομεί που θα εξαιρεθούν από το σύστημα εμπορία, να πω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Όλες αυτές οι εγκαταστέσεις καλύπτονται από το σύστημα εμπορία. Και επειδή ένα τομέα ή υποτομέα βρίσκεται στον κατάλογο διαρροή άνθρακο, δεν θα καλύπτεται από το σύστημα εμπορία θα καλύπτεται ακόμα και αν παίρνουν 100% ε, άδεια αυτό με βάση μια συγκριτική μελέτη αποτελεσματικότητας. Ε, που ορίστηκε ανάμεσα στο ε, Κοινοβούλιο Συμβούλιο πέρυσι με πολύ αυστηρό επίπεδο. Από του χρόνου θα οριστούν τα συγκεκριμένα επίπεδα και για κάθε τομέα και υποτομέα πρέπει να βρισκόμαστε γύρω στο μέσο όρο ε, των βέλτιστων αποτελεσμάτων, του 10% των βέλτιστων αποτελεσμάτων στους τομείς και στου υποτομείς. Και μόνο οι εγκαταστάσει που βρίσκονται στο επίπεδο αυτό θα έχουν όλε τι ποσοστώσεις δωρεάν. Οι άλλοι θα πρέπει να αγοράσουν, είτε απευθείας, είτε στη δευτερογενή αγορά. Αυτά ήθελα να πω και να τα θυμάστε. Ευχαριστώ. Πράγματι ήταν σημαντική αυτή η διαπίστωση καθώς υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις. Λοιπόν, κύριε κυρία Ρογανά, πλάμπ τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τα σχόλια της ε, Κομισιόν. Θα ήθελα εγώ να χαιρετήσω την συνεισφορά της ε, Κομισιόν και συγκεκριμένα το σημείο αυτό που είπε πως πρέπει να έχουμε μια οικονομία η οποία θα εξελίσσεται συνεχώς, θα κινηθεί σε μια πράσινη κατεύθυνση και αν θέλουμε βεβαίω να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας δεν θα πρέπει να εισαχθούν εδώ πέρα στοιχεία διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τους κλάδους της βιομηχανίας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως κάποιοι κλάδοι πρέπει να μελετηθούν ακόμη μία φορά όσον αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών. καθώς επίσης και ο τομέας των πλακιδίων καθώς βεβαίως σε όλες τις οικοδομές ε, ε, χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται και στο μέλλον ε, αυτός ο τομέας. Τώρα η απάντηση της Κομισιόν σε σχέση με τα δεδομένα από αυτόν τον τομέα που έχουν φτάσει στην Κομισιόν, τα οποία δεν τα πιστεύουν γιατί δεν είναι από επίσημες πηγές, είναι κάτι που δεν το αντιλαμβάνομαι. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να ξαναμελετήσει αυτόν τον τομέα, όχι μόνο για τη Ρουμανία, ε, γιατί είναι σημαντικό βεβαίως αυτό και για τη χώρα την οποία εκπροσωπώ, αλλά και για τις άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ, Λίντα Μάγκεν. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούω μερικούς να λένε ότι το να έχουμε τον κατάλογο ήδη έτοιμο πριν από την Κομπεχάγη δυσκολεύει τη διαπραγματευτική μας εντολή. Αλλά το αποφασίσαμε αυτό ήδη πέρσι στην νομοθετική διαδικασία, βάσει της οποίας η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη μέχρι το τέλος του 2009, 10 λέει η ομίλητρια, να έχει αυτόν τον κατάλογο. Νομίζω ότι το Συμβούλιο δέχτηκε το τέλος του 2010 και επομένω η Κομισιόν υποχρεωμένη να έχει αυτό το κατάλογο μέχρι το τέλο του 2010 βάσει τη νομοθεσία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη συμφωνία. Εγώ έχω αντιμετωπίσει πιέσεις και από τη βιομηχανία και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να αλλάξουμε αυτό τον κατάλογο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον αλλάξουμε. Ό,τι αποφασίστη, απεφασίστη. Και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο δημιούργησε πολλά προβλήματα για βουλευτές του Κοινοβουλίου μερικοί θέλαν αυτόν τον κατάλογο να τον έχουμε ακόμα νωρίτερα. Πρέπει τώρα να μας πει η Κομισιόν. Αυτό θα μας δημιουργήσει προβλήματα στη διαπραγματεύση. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες δημιουργούν, δημιουργούν τους δικούς τους καταλόγους για τις διαπραγματεύσεις. Ορισμένοι ζητήσανε να αυξήσουμε τις, ε, τις να, μάλλον να, να φέρουμε το κατάλογο να ισχύει μέχρι το 20, 2020, ενώ εμείς έχουμε πρόβλεψη μόνο μέχρι το 2014. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα προκύψει μετά το 2014, ούτε θέλουμε να προσθέσουμε τομείς. Ήδη είναι πάρα πολύ μακροσκελής ο κατάλογος. Πολλοί θέλουν να είναι πιο περιορισμένος ο κατάλογος. Πολλοί θέλαν να καταλογίζεται, να καταγραφεί και το έμεσο κόστος στον κατάλογο. Πολλοί τομείς βρίσκονται εδώ γιατί προσθέσαμε και κριτήρια πέρσι σε σχέση με τα οποία τα κριτήρια σε σχέση με τα οποία η Κομισιόν θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, η Κομισιόν βρίσκεται απόλυτα μέσα στα πλαίσια της εντολής της. Άκουσα τι εξηγήσει της για τον αντίκτυπο σε τρίτες χώρες. Αν γίνει λοιπόν αυτή η αξιολόγηση στην Κοπενχάγη, εγώ δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση των τρίτων χωρών πριν από την Κοπενχάγη. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο κατάλογο πραγματικά θα πρέπει να καταρτιστεί στα μέσα του επόμενου χρόνου αυτό θα ήταν πιο επωφελές. <clears throat> Προς το παρόν λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι η Κομισιόν έκανε ό,τι της ζητήσαμε μέσα στα πλαίσια αυτού του νομοθετήματος. Ευχαριστώ. Και ο Ρίχαρτ τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μακροσκελισμένο κατάλογος, αλλά θα πρέπει να είναι και μακροσκελής Και σίγουρα ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε και την ε, ε, αποδοτικότητα της ενέργειας. Στην Ευρώπη είναι διπλάσια αυτή η αποδοτικότητα ενέργειας από χώρες οι οποίες δεν έχουν προβεί σε αντίστοιχες προσπάθειες στον τομέα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι και η Κομισιόν έχει δυνατότητα, πρέπει να εξασφαλίσουμε το κατάλογο αυτό, την δυνατότητα της Ευρώπης να συνεχίζει να παράγει. Αυτό το οποίο τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μια έλλειψη διαφάνεια στη διαδικασία αυτής της διαδικασίας. Το Κοινοβούλιο γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι ικανοποιημένο με την επιτροπολογία, τη διαδικασία λήψη απόφασης για την τροποποίηση των κανόνων. Θα ήθελα όμως να ξέρω η Κομισιόν βάσει ποιων αρχών, ποιων κριτηρίων προχωρά για την ε, κατάρτιση του καταλόγου και ίσως θα έπρεπε να βελτιώσει την παρουσίαση κατά και επιμέρους τομείς. Εμείς έχουμε ένα σύστημα εδώ το οποίο έχει τεράστιες επιπτώσεις σε οικονομικό και βιομηχανικό τομέα για όλη την Ευρώπη. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν νομίζω ότι ορθά παρέπεμψε στη διαδικασία του benchmarking. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία από την πλευρά της Κομισιόν να εξηγήσει ότι οι φορείς αυτής έχουν ε, υποβάλλονται στη διαδικασία του benchmarking, αλλά θα έπρεπε η Κομισιόν επίσης να μας πει πώς προβλέπει σε συγκεκριμένο επίπεδο να εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία του benchmarking και ποια είναι η, η προβλεπόμενη συμμετοχή του Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σημείωσα τις παρεμβάσεις ε, που αφορούν τον τομέα των ε, της πληθοποίας και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο ε, ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ορισμένα κράτη-μέλη και στην ε, διαδικασία επιτροπολογίας με τα κράτη-μέλη προσθέθηκε μια νέα σκέψη στην πρώτη επιτροπή σύμφωνα με την οποία ε, καλεί το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναξιολογήσει το τομέα αυτό στον τον πιο γρήγορα. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. ανέφερα επίσης και ε, άλλους ε, τομείς που θα εξεταστούν. Ε, σίγουρα πάντως θα τα κάνουμε αυτά μέσα στους επόμενους μήνες. Συναντηθήκαμε με, το, με σε εκπροσώπους του τομέα για να μπορέσουμε να δούμε τι στοιχεία θα πρέπει να παίρνουμε ε, και, να το, και θα ελέγξουμε τα αποτελέσματα αυτά και με τα κρατημέλη. Θα γίνουν λοιπόν όλα αυτά. Ευχαριστώ την κυρία Μακέβαν γιατί μας υπενθύμησε την νομοθεσία και το τι ακριβώς αναφέρει. Στην ουσία βεβαίως δεσμευόμαστε ε, από, και από την νομική προθεσμία προς το τέλος του χρόνου και από μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θεωρήσαμε ότι αυτή ήταν η σωστή προσέγγιση δεν υποβάλαμε την πρόταση και διαφωνήσαμε και στη διαδικασία στην απόφαση, αλλά το αποφάσισαν οι σύνομοθέτε. Άρα τουλάχιστον αυτό το χρόνο με την, ε, με την ενθεώρηση μετά την Κομεχάγη, αυτά θα πρέπει να δώσουμε. Βεβαίω, παίρνουμε ερωτήσει από τι τρίτε χώρε, γιατί είδαν το σχέδιο καταλόγου, δεν εγκρίθηκε επίσημα. Θέλουμε πρώτα ε, τη δική σα εξέταση και την επιβεβαίωση του Συμβουλίου τη ψήφου από τα κράτη-μέλη και μετά επίσημη έγκριση από την Επιτροπή το Δεκέμβριο. Πάντω, παίρνουμε ερωτήματα. Και το γεγονό ότι ακολουθήσαμε μια ιδιαίτερα στοχοθετημένη ε, και αναϋποτομέα ε, ε, προσέγγιση, είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μακροσκελή κατάλογα Αλλά επειδή έχουμε πολλούς υποτομείς, αν ακολουθούσαμε ένα υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης, θα καλύπτουμε τις ίδιες εκπομπές, ακόμη και περισσότερες, αλλά θα είχαμε λιγότερους τομείς. Εδώ όμως θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε και να εντοπίσουμε συγκεκριμένους τους υποτομείς. Έχουμε πολλά ερωτήματα και πρέπει να δώσουμε πολλές εξηγήσεις, βεβαίως. Το γεγονό λέει ότι βρίσκεται κανεί στον κατάλογο δεν εξαιρείται από το σύστημα, το αντίθετο. Τίθεται ερωτήματα. Δεν μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή ότι έχει δημιουργήσει πολλή αναταραχή μέχρι αυτό το στάδιο, αλλά σίγουρα έχει, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ε, ήδη ε, αναφέρθηκαν, αναφέρθηκε το θέμα των τούβλων και επίση όσον αφορά τον κύριο Ζήμπερ και αυτά που είπε για περισσότερη διαφάνεια και συμμετοχή των εμπλεκομένων και των ενδιαφερομένων. Από τότε που αρχίσαμε την ανθεώρηση ε, του συστήματο εμπορία. Ε, στόχος ήταν πλήρης διαφάνεια και πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Και σε κάθε συνεδρίασή μα για το θέμα τη διαρροή του άνθρακα έρχονται οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων. Και στα πλαίσια τη συναπόφαση είχαμε τρει ή τέσσερι συνεδριάσει τουλάχιστον πριν από την ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, το Σεπτέμβρη. Είχαμε πολλέ ε, πολυμερεί ε, συναντήσει ε, με όλου. Ε, υπήρχαν ερωτήσει για τη μεθοδολογία. Σα παραπέμπω στην αξιολόγηση αντικτύπου, όπου έχουμε πλήρη περιγραφή τη μεθοδολογία, ε, του τρόπου υπολογισμού του κόστου κτλ. Όλε αυτέ οι πληροφορίε βρίσκονται και στην ιστοσελίδα μα. Να σας το ξαναπούμε, στο σελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και έχουμε συνεργαστεί μαζί τους πολύ. Αν δεν είχαμε τα δικά του στοιχεία, το πιο πιθανό να μην είχαμε τον κατάλογο με τη σημερινή του μορφή. Επίσης, όσον αφορά ε, τις, ε, ε τα συγκριτικά επίπεδα, ήδη είχαμε ορισμένες συνεδριάσεις με τους ενδιαφερομένους, γιατί θα κάνουμε προς την κατεύθυνση των benchmarks. Ε, συνεργαζόμαστε με τους συμβούλους προς την κατεύθυνση αυτή, που θα ολοκληρώσουν την πρώτη τους έκθεση, εξετάζοντας τις βέλτιστες επιδόσεις και το 10% των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε διατομείς και υποτομείς και ε, τις τιμές των εκπομπών για τους αντίστοιχους υποτομείς. Ε, θα το έχουμε στι επόμενες προσεχείς εβδομάδες και μετά θα μπούμε στο δεύτερο επίπεδο συζητήσεων αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε δεύτερη συνάντηση και εκεί ε, και μέσα στου επόμενου μήνε θα έχουμε και άλλε τέτοιε συνεδριάσει για να προετοιμάσουμε την πρόταση τη Επιτροπή πριν από το καλοκαίρι και μετά τη διαδικασία απόφαση, όπω ακριβώ και στον κατάλογο ε, για τη διαρροή του άνθρακα, ε, του ε, τελευταίου μήνε του 2010. Πλήρη επικοινωνία λοιπόν με του ενδιαφερομένου. Το κάναμε ήδη. Βεβαίω σήμερα δεν μπορούμε να δώσουμε όλε τι λεπτομέρειε για το πώ ε, θα καταλήξουμε σε συγκριτικά επίπεδα αναφορά. Πρέπει να το συζητήσουμε με του εκπροσώπου του κλάδου, με του ενδιαφερόμενου. Δεν μπορούμε να σα δώσουμε λεπτομέρειε περισσότερε τώρα. Έχουμε άλλο ένα χρόνο στη διάθεσή μα για να εργαστούμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τον επόμενο κύριο, ο Καρλ Χάιντ Φλόρεντ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, κατα... στην συζήτηση για αυτό τον κατάλογο πρέπει να σκεφτούμε ποιες αρμοδιότητες έχουμε εμείς και να επικεντρωθούμε στο, στο έγγραφο που έχουμε τώρα μπροστά μας. Βεβαίω, υπάρχουν πολλές ιδέες που μπορούμε να συζητήσουμε για όλο το ζηματιοξίδιο του άνθρακα. Αλλά εγώ θα συμβούλευα σε αυτό εδώ το έγγραφο να συγκεντρωθούμε, να πούμε ένα ναι και να φυλάξουμε το μπαρούτι μας, αν θέλετε, τα πυρομαχικά μας για το επόμενο έγγραφο που θα μας έρθει εκεί πέρα πράγματι ο χώρος ε, ελιγμών της ε, Κομισιόν είναι πολύ μεγαλύτερος για να απογκριθούμε από τις ε, πολιτικές ιδέες που υπάρχουν. Κοίταξε, τέλειος δεν θα είναι ποτέ αυτός ο κατάλογος. Θεωρώ πως έχουμε λοιπόν περισσότερο χώρο λιγμών στα benchmarks. Οπότε πρέπει να τα αποδεχτούμε τώρα τα πράγματα όπως έχουν. Βεβαίως μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα τι γίνεται πως έχουμε φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί εμείς μιλήσαμε για 100%, μετά μας είπαν και το 80% μια χαρά νούμερο είναι και μετά φτάσαμε στο 75%. Φαντάζομαι η Κομισιόν θα μας ε, εξηγήσει τέλος ή να τα εξήγησε μπορεί, δεν ξέρω εγώ έλειπα και στην αρχή και ζητώ συγγνώμη. Θεωρώ πως εδώ πέρα όπως έχουν τα πράγματα και όπως έχει και η νομοθεσία εντάξει, με κάποια δυσκολία μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά σας παρακαλώ να φυλάξουμε την, την δύναμή μας και στους άλλους δύο φακέλους εκεί να εξαντλήσουμε την ε, κοινοβουλευτική μας ε, δύναμη. Βεβαίως ε, το θέμα των benchmarks μπορούμε να το ερμηνεύσουμε τελείως διαφορετικά προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση και μπορούμε να επικεντρωθούμε π.χ. σε μία χώρα μόνο και να το ή να το οργανώσουμε ίσως σε μια χώρα και να το συζητήσουμε σε μια ωραία χώρα, ελπίζω. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να κάνω μία προσωπική παρατηρήση. Βλέπω εδώ πέρα και την εισηγήτρια. Και όσον αφορά το ε, θέμα του συστήματος εμπορίας εκπομπών, έχουμε τσακωθεί βέβαια πάρα πολύ, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που την βλέπω. Α, βλέπω πως τελικά υπάρχει μία συμφιλίωση στο τέλος. Απορώ πως δεν είναι σαν του χάσει στο, στον κατάλογο μου. Ε, επειδή σήκωσε λοιπόν τελικά το, το καρτελάκι, είναι και στον κατάλογο. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ που με είδατε, τα ανέβματα που έκανα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον, τους εκπροσώπους της Κομισιόν για τις απαντήσεις οι οποίες έχουν διαλευκάνει πάρα πολλά θέματα και επίσης ε, για τους συναδέλφους οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα. Υπάρχουν ε, νομικά θέματα, υπάρχουν οικονομικά θέματα και υπάρχουν και θέματα διεθνούς χαρακτήρα. Η Λίντα Μακρύβαν, όπως και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν, είπαν ότι η καταληκτική προθεσμία ότι οι χρονικές διαδικασίες έχουν καθοριστεί από το νομοθέτημα το ίδιο. Κάτι όμως το οποίο δεν έχει ληφθεί υπόψη από την Κομισιόν, από την Κομισιόν στις αξιολογήσεις της είναι το άρθρο 10 παράγραφος 18 για τις τρίτες χώρες και τα κριτήρια των τρίτων χωρών. Εκεί λέει το νομοθέτημα ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη δράση των τρίτων χωρών και τον βαθμό στον οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα των άλλων χωρών για την κλιματική αλλαγή. Και φυσικά ο βαθμός στον οποίο τα μέτρα αυτά είναι συγκρίσιμα με τα δικά μας. Εγώ πληροφορήθηκα ότι η χαλιβουργία της Βραζιλίας έχει μία αποδοτικότητα ο τομέας αυτός που είναι εξίσου υψηλή με της Ευρωπαϊκή χαλιβουργίες. Τέτοια θέματα δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην ε, αξιολόγηση στην οποία προέβη η Κομισιόν. Επομένως, τα κριτήρια του νομοθετήματος δεν έχουν ακολουθηθεί πλήρως. Και υπάρχει ένα ερώτημα ένα πρόδειλο ερώτημα το οποίο έλκεται από όλα αυτά. Τι προβλέπει να κάνει λοιπόν, τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν. Μπορεί το θέμα αυτό να ληφθεί υπόψη όταν εσείς κάνετε μία εκτίμηση όταν αντιμετωπίζετε, όταν προσπαθείτε να καθορίσετε την ένταση εμπορίου στον τομέα αυτό. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι το εμπόριο με τις χώρες αυτές όπου τα μέτρα για την αποτελεσματικότητα της βιομηχανίας ό,τι αφορά τη χρήση της ενέργειας και τα κλιματικά μέτρα όταν είναι παρόμοια αυτά τα μέτρα με τα δικά μας, τις αποκλείεται αυτές από την εξέταση της έντασης εμπορίου. και άλλα δύο σχόλια γενικού χαρακτήρα. Για το γιατί πιστεύω ότι απέχει παρασάγκας αυτή η, αυτό το, αυτή η νομοθεσία από αυτό το οποίο είναι απαραίτητο. Υπάρχει καταρχήν ένα θέμα οικονομικό. Στην ακρόαση που οργάνωσε η κυρία Ντόιλ το προηγούμενο έτος, μας ελέγχθη ότι δεν είναι βέλτιστη, βέλτιστα κατά 100% τα εναλλακτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά η εναλλακτική λύση θα ήταν όχι δωρεάν παροχή, αλλά πλή, πλήρης δημοπράτηση και μέτρα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δωρεάν παροχή εκπομπών σημαίνει ότι οι βιομηχανίες οι οποίες έχουν αυτήν την ε, ε, άδεια εκπομπής μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές τους και να, δώσουν, να τα πουλήσουν σε άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη λεγόμενη διαρροή άνθρακος. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή το μήνυμα το οποίο δίνουμε στον διεθνή χώρο πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Διάβασα, ίσως και άλλοι διάβασαν, συνάδελφοι, τη διαδικασία για την ε, κλιματική νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναφέρεται το επιχείρημα ότι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία φαίνεται να υπάρχει και η υπόσχεση μιας δωρεάν κατανομής εκπομπών και αυτό το χρησιμοποιούν οι νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι αγωνίζονται να πετύχουν την καλύτερη δυνατή νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και μας λένε ότι οι Ευρωπαίοι μας δυσκολεύουν τη ζωή μας. Είναι δύσκολο για μας να υποστηρίξουμε πιο αυστηρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος όταν οι Ευρωπαίοι είναι ανοιχτοχέριδες και προτείνουν 100% δωρεάν παροχή εκπομπών στις βιομηχανίες. Πολύ ωραία. τι είναι. Ευχαριστώ. Όλοι ξέρουμε τι θα προκύψει λοιπόν αυτή τη στιγμή στην Κοπενχάγη. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει τώρα για την κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα ενέργειας για όλους τους τομείς της βιομηχανίας. η Κομισιόν θα πρέπει να αξιολογήσει και τις δράσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα σε χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτού καθοριστεί ο οριστικός κατάλογος τομέων. Γι' αυτό εγώ δεν νιώθω πολύ καλά με την πρόταση αυτή. Γιατί εγώ δεν βλέπω να υπάρχει μια τέτοια επιστημονικο-οικονομική ανάλυση η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει το να θέσουμε τόσο χαμηλά τα κατόφλια, όπως κάνει η Κομισιόν. Και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να, είχα, να έχω περισσότερη διευκρίνηση από την πλευρά της Κομισιόν. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ο Κομισιόν βασιπίων πηγών, βασιπίων δεδομένων για τρίτες χώρες σε σχέση με την αποδοτικότητα χρήσης ενέργειας στις τρίτες χώρες και σε, έχουν βασιστεί και σε ποιες περιπτώσεις ήταν αδύνατο να προβείται σε μια αξιολόγηση λόγω ελλείψεως δεδομένων. Μήπως θα μπορούσατε επίσης να μας δώσετε και περισσότερα στοιχεία και να τα δημοσιεύσετε εξάλλου την μεθοδολογία βάσει της οποίας προσπαθήσατε να αξιολογήσετε όλα αυτά τα στοιχεία και ποια είναι τα σχέδιά σας για να έχετε μια πληρέστερη αξιολόγηση που να έχει μεγαλύτερη κάλυψη. Επίσης θα ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν αν ζήτησε δεδομένα από τρίτες χώρες για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας χρήσης ενέργειας και των αποτελεσμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο από τρίτες χώρες. Κατά πόσο λοιπόν όλα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Κομισιόν, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ δυσάρεστα με αυτή την πρόταση. Νομίζω είναι απλώς πολύ χαμηλά τα επίπεδα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με χρονολογική σειρά. Το ερώτημα του κυρίου Φλόρεντς για τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν μίλησε ότι ξεκινήσαμε από ένα 100% που κατέληξε τελικά στο 75%. Η πρόταση της ε, δηλαδή. Αυτό έγινε μετά από στενή συνεννόηση με την νομική υπηρεσία γιατί αναγκαστήκαμε να κοιτάξουμε πάρα πολύ ε, λεπτομερό τον ορισμό του κόστου στο άρθρο 10α παράγραφο 15 όπου λέει πω πρέπει να εξετάσουμε το επιπλέον κόστο που προκύπτει από την εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Εάν λάβετε υπόψη πω ο κατάλογο θα ισχύσει μόνο για 5 χρόνια και θα υιοθετηθεί το τέλος 2009, οπότε θα είναι μέχρι το τέλος 2014. Έχουμε λοιπόν δύο έτη, το 2013 και 2014 της τρίτης φάσης εμπορίας που θα καλυφθούν. Το ε, κανονικό επίπεδο σε αυτά τα δύο έτη θα είναι 80% και μετά θα πέσει κατά τη διάρκεια των ετών. Οπότε έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το επίπεδο των δωρεάν ε, αδειών εκπομπών και το τι νομίζουμε ότι θα προκύψει από τη συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά την αυστηριότητα και μιλάμε για ένα αρκετά αυστηρό αποτέλεσμα. Δηλαδή μόνο οι καταστάσεις οι οποίες είναι μόνο στο κορυφαίο επίπεδο αποτελεσματικότητας θα λάβουν 100% άδειες. Εάν, προστα... πολλαπλασιάσουμε αυτούς τους δύο παράγοντες μιλάμε για 75% δημοπράτηση που πρέπει να είναι λογικά το κανονικό σενάριο για όλε τι εγκαταστάσει και ήταν σαφή η νομική μα υπηρεσία. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση και πάμε στο 100% θα μπορεί να προσβληθεί πολύ εύκολα η απόφαση νομικά, κάτι το οποίο δεν συμφέρει ούτε βιομηχανία να έχουμε μια απόφαση η οποία θεωρούν ότι είναι νομικά βέβαια, αλλά μετά προσβάλλεται πολύ εύκολα για την ανάλυση των τρίτων χωρών. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό πράγματι. Προσλάβαμε και συμβούλους, να δούμε τι δεδομένα υπάρχουν. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο, τα δεδομένα που υπάρχουν είναι ad hoc, δεν είναι συγκρίσιμα. Επίσης, ε, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως ναι, πράγματι υπάρχουν πολλά υποσχόμενες εξελίξεις σε πολλές τρίτες χώρες, αλλά ποιε τρίτες χώρες έχουν νομοθεσία πού είναι νομικά δεσμευτικέ αυτές οι προσπάθειες. Ξέρουμε πως η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν ε, καλύπτονται από το ευρωπαϊκό σύστημα μέσω του ΕΟΧ και η Ελβετία έχει κάποια νομοθεσία, αλλά πέρα από αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια ανάλογη δέσμευση η οποία να είναι νομικά δεσμευτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το ξαναδούμε το ζήτημα μετά την Κομεχάγη, γιατί οπωσδήποτε όπω και εσεί έτσι και εμεί ελπίζουμε πω μετά την Κομεχάγη θα είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για το ποιε είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν αυτέ οι χώρε και το εάν θα τι εφαρμόσουν. Όπως είπα, χρησιμοποιούμε συμβούλους, δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, αλλά την αναμένουμε τις ερχόμενες εβδομάδες και βεβαίως ε, θα γίνει διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα μας, αλλά είναι ένα ζήτημα που θα το παρακολουθήσουμε και είναι ένα σημαντικό στοιχείο μετά την Κομεχάγη. Και αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Χάση, για να κοιτάξουμε τα δεδομένα του εμπορίου θα δούμε το τι κάνουν οι τρίτε χώρε και θα το ενσωματώσουμε στην αξιολόγηση των εμπορικών δεδομένων. Η κυρία Κάνεν ανέφερε επίση το γεγονό πω ε, το ποσοστά ε, είναι πολύ χαμηλά. Πράγματι, αυτό το συζητήσαμε κατά τη διάρκεια τη συναπόφαση πέρσι και αυτό προέκυψε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, σε αυτό βασιζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αφείς ε, απαντήσεις. Ε, θα ήθελα όμως μια διευκρίνηση ακόμα. το ΜΕΑΣ τον ανέφεραν αρκετοί συνάδελφοι. Ακούω πως υπάρχουν εδώ πέρα πολλοί υποστηρικτές ε, των τούβλων και των πλακιδίων. Η Κομισιόν λέει ναι, το κοιτάμε, θέμε προφορίες, θα γίνει το συντομότερο δυνατόν και τους ερχόμενους μήνες το ερώτημά μου συγκεκριμένα είναι θα το καταφέρετε τους ερχόμενους μήνες πριν το τέλος του έτους. Γιατί καλό θα ήταν να έχουμε και για αυτόν τον τομέα συγκρίσιμα στοιχεία ταυτόχρονα με τους άλλους τομείς. Ή περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κάτι συγκεκριμένο του χρόνου και να πάει στην ε, αναθεώρηση, δηλαδή να καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τελικά ως αποτέλεσμα. Αυτή είναι η απάντηση που θέλω. Uh, Κοιτάξτε, τα πραγματικά προβλήματα, όπως είπε η κυρία Μακέβανς, ε, ε, είναι, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η νομοθεσία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Είναι παράξενο, για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχουμε 100% δωρεάν μόλις κανείς πλήρει τα κριτήρια. Ίσως θα έπρεπε να το 100% αυτό να οφείλεται, ε, να, να αποδίδεται στις εκπομπές πάνω από τα κριτήρια. Ε, αυτό θα ήταν πιο λογικό. Αλλά μόλις κανείς πληρεί τα κριτήρια τότε 100% δωρεάν. Ε, αυτό παράξενο. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να αναφερθώ στα συγκριτικά επίπεδα αναφοράς. Γιατί μπορείτε να τα επηρεάσετε, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κανονισμό. Λέτε Το 2007-2008 είναι το έτος προσδιορισμού αυτών των επέδων. αλλά θα εφαρμοστούν και το 2013-2014. Άρα δεν έχετε ε, κριτήρια αιτήσεις αποτελεσματικότητας. Και αυτοί που είχαν τις 10 καλύτερες επιδόσεις 2007-2008 ε, και το 2013-2013, γιατί αν έχουμε ε, ένα διαφορετικό συντελεστή αποτελεσματικότητας, τότε ε, θα μειωθούν τα επίπεδα αυτά. Αν έχουμε 1,5. Αν όμως έχουμε 2,5 δίκτυα αποτελεσματικότητα που έχουν ορισμένοι από αυτού. τότε θα έχουμε 14% μείωση αυτού του συγκριτικού επίπεδου. Θα λάβετε υπόψη ε, τον ετήσιο δίκτυο αποτελεσματικότητας και θα κάνετε αναγωγή για το 2014, 2013-2014. Διαφορετικά δεν θα έχετε σωστά αποτελέσματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ο Έκοτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπαμε πολλά για τις αδυναμίες του νομοθετήματος. Το ξέρω, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι μέσα σε αυτό το νομοθέτημα να προσθέσουμε στον κατάλογο αυτό κάθε χρόνο τομείς και εταιρείε. Αλλά για να τις βγάλουμε από τον κατάλογο αυτό μπορεί να γίνει μονάχα μια φορά που είναι αυτή η διαδικασία αναθεώρησης μετά την Κομπεχάη. Ας δώσουμε λοιπόν πιο πολύ βάση σε αυτή τη διαδικασία και ας έχουμε σαφείς απαντήσεις από την Κομισιόν. Πότε ακριβώς θα γίνει αυτή η αναθεώρηση του καταλόγου και εξετάζεται κάτι το οποίο εγώ θα σας συνιστούσα να προσαρμόσετε τους υπολογισμούς του έμεσου κόστους γιατί αυτή τη στιγμή βασίζονται σε μέσο όρο εκπομπών που δεν είναι η σωστή βάση. Και στη συνέχεια το επόμενο ερώτημα είναι πότε προβλέπει η Κομισιόν θα έχει καλύτερα στοιχεία από τις δύο χώρες για την αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας ώστε να χρησιμοποιήσει αυτό το κριτήριο στην αναθεώρηση, γιατί είναι κριτήριο που βρίσκεται στην νομοθεσία, δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τον τρέχοντα καν κατάλογο, αλλά να χρησιμοποιηθεί στον αναθεωρημένο κατάλογο, ώστε να ξέρουμε ότι έχουμε τις σωστές εταιρείε σε αυτόν τον κατάλογο. Κυρία Σλίμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τα τούβλα. Θα τα κοιτάξουμε τα τούβλα. Και είχαμε μια συνάντηση με τους αρμόδιους κλάδους. Βάσει των στοιχείων που έχουμε, ο επιμέρους αυτός τομέας δεν καλύπτει τα κριτήρια. Αν λοιπόν ε, ένα τομέα ή κάποιο κράτος μέλος μπορεί να, θέλει να επιχειρηματολογήσει ότι ο τομέας των τούβλων θα εκτεθεί σε διαρροή άνθρακος, θα πρέπει να παρουσιάσουν νέα στοιχεία. Εναπόκειται λοιπόν στον τομέα ή σε ένα κράτο μέλο να κάνει αυτή την επιχειρηματολογία. Εμεί δεν μπορούμε λοιπόν να δεσμευτούμε. Εξαρτάται από το πότε θα μα δοθούν τα στοιχεία και θα τα εξετάσουμε το ταχύτερο δυνατό. Αλλά πρέπει να είμαστε σαφεί ότι ο τομέα αυτό δεν θα προσθεθεί στον τρέχοντα κατάλογο. Δεν μπορεί γιατί εξάλλου και τούβλα. Αν γίνει λοιπόν αυτή η αλλαγή στον κατάλογο, θα πρέπει να υπάρξει και πάλι έγκριση από τα κράτη-μέλη και αυτό σημαίνει θα χάσουμε την καταληκτική προθεσμία για το τέλος του χρόνου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, μπορούν να προσθεθούν νέες εταιρείε και νέοι τομείς στην επόμενη αναθεώρηση που δεν πρέπει να γίνει μονάχα του χρόνου, αλλά και τα επερχόμενα έτη και μπορεί η Κομισιόν να προσθέσει στον κατάλογο. Για το ερώτημα του κ. Σλίχτορ για την διαδικασία του benchmarking, της βαθμονόμηση. αυτό είναι εν εξελίξη. Σίγουρα δεν περιμένετε να σας δώσω τις πλήρες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό εδώ και τώρα. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι τα σημεία εκκίνησης του benchmarking έχουν καθοριστεί σαφώς στην νομοθεσία και η Κομισιόν θα πρέπει να βασιστεί στις παραμέτρους που αναφέρονται στο νομοθέτημα που είναι ο μέσος όρος του καλύτερου 10% για κάθε τομέα και για κάθε υποτομέα. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία αναφέρονται που είναι τεχνολογική ανάπτυξη, ικανότητα αντικατάσταση κτλ. Και θα τα εξετάσουμε και αυτά. Για τη δεύτερη φάση έχουμε επίσης την πρόβληση του benchmarking, πραγματικά για εγκαταστάσεις παραγωγής ε, λιπασμάτων, όπου υπάρχουν ε, ήδη κάποια benchmark από την Αυστρία ή τις κάτω χώρες και έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατεβαίνουν κάθε χρόνο τα benchmark. Και αυτό είναι δυνατό αλλά ακόμα και αν έχετε ένα συγκεκριμένο benchmark το οποίο θα εφαρμόσετε σε μια χρονική περίοδο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει η ετήσια μείωση κατά 1,74% στο συνολικό επίπεδο εκπομπών που περιλαμβάνει και το benchmark, περιλαμβάνει και τις δωρεάν εκπομπές, 1,74 κατεβαίνει κάθε χρόνο. Οπότε πάντα έχουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι ποσοστό απομείωση. Εάν όμω επί τη βάση των ιστορικών δεδομένων παραγωγή εξακολουθεί να είναι 100% και βάσει του benchmark θα ξεπερνούσαμε το επίπεδο το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία, προβλέπεται και ένα παράγων, ένα συντελεστή διόρθωση. Όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνουν και την δυνατότητα να μειωθεί σε σχέση με το benchmarking, κάτι το οποίο είναι υπερβολικά γενναιόδρος. Αυτά που λέει ο κύριος Eckhout η Κομισιόν έχει την εντολή να καταλήξει με μια έκθεση μέχρι τον Ιούλιο, Ιούνιο του 2010 που να περιλαμβάνει και τα συμπερασμάτια της Κοπενχάγης και θα πρέπει να δούμε τότε μετά τι μας δίνει αυτή η αξιολόγηση για να δούμε τι θα κάνουμε εάν προχωρήσουμε σε αυτή την ε, προσέγγιση για τη διαρροή άνθρακος, αν πρέπει να αλλάξουμε τον κατάλογο, όλα μπορούν να γίνουν στην Κοπεχάγη, καλά αποτελέσματα, κακά αποτελέσματα, 20% μπορεί να φτάσουμε στο 30%. Γενικά λοιπόν δεν μπορώ σήμερα να σας πω τι θα γίνει. Ποια θα είναι η κατάσταση μετά την Κοπεχάγη. Όπως σας είπα, μετά από την Κοπεχάγη θα επανεξετάσουμε το θέμα των τρίτων χωρών, των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τρίτες χώρες, αν τις εφαρμόζουν με νομικά δεσμευτικό τρόπο, αν θα είναι νομικά δεσμευτικό το αποτέλεσμα της Κοπεχάγης και αυτό είναι ένα ερώτημα άξιων απαντήσεως και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, δράση μας. Θα έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να το πράξουμε. Θα σας δώσουμε λοιπόν τη μελέτη όταν την έχουμε και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε δεδομένα για τις τρίτες χώρες και τη συγκεκριμένη την ε, συγκρισιμότητα των δεδομένων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο για την αναθεώρηση που έχει να κάνει με το, μετά την Κοπενχάγη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ εκ βάθους καρδίας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος θα αναλάβει λάβει το λόγο. Είναι ένα απαράγραπτο το κομμάτι του συστήματος κλιματικής, αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και επομένως θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να το εξετάζουμε. Ακούσαμε από την κυρία Λίνσπερ και την Κομισιόν ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Την ευχαριστώ. Προθεσμία τροπολογιών 8 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι το μεσημέρι τη 8 Οκτωβρίου λοιπόν μπορούν να κατατεθούν τροπολογιε Η επόμενη συνεδρίαση μας 19 Οκτωβρίου, Δευτέρα, το βράδυ στο Στρασβούργο θα ψηφίσουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το κλιματική αλλαγή πέρα συνεδρίαση.